morbidity and mortality να εμφανιστεί ω υποστηρικτής και αξιολογητής της εναλλακτική ε, διευθέτησης διαφορών και όχι ω φορέα που θα την επιβάλλει υποχρεωτικά. Να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί να ανθίσει με τον δικό της τρόπο εναλλακτική διευθέτηση διαφορών. Βέβαια αυτό μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο. Αν θέλουμε ωστόσο η ενιαία αγορά να επωφεληθεί από την αλλακτική διευθέτηση διαφορών, αυτό είναι ο σωστό δρόμο. Σα ευχαριστώ. Uh, well, thank you very much indeed, Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις πολύ εύστοχες αυτές οι ιδέες εν εκτροπή μου μετέβηε στην συμβολή στη συζήτηση και νομίζω ότι ήταν και πολύ πρακτικέ ε, οι σύμβουλε αυτέ από κάποιον ο οποίο έχει εργαστεί στον κλάδο. Και όταν πρόσφατα, όταν η Επιτροπή μου μετέβη στην Ουγγαρία, χαρήκαμε που γνωρίσαμε τι σχετικέ αρχέ προστασία του καταναλωτή στην Ουγγαρία και συζητήσαμε το έργο του. Να συνεχίσουμε τώρα τι παρουσιάσεις μας και είμαι πολύ περήφανος ε, που έχουμε μαζί μας την Πάολα Τεστορικότζη ως ε, υπεύθυνη του σχεδίου αυτού για να μας μιλήσει. Ευχαριστώ Μάλκολμ και να σας ευχαριστήσω ως πρόεδρο της Επιτροπής ΙΜΚΟ για την υποστήριξή σας ε, για το θέμα αυτό για μας από πλευράς ε, πολιτικής καταναλωτή. Ήταν πάντα πολύ σημαντική η εναλλακτική μέθοδη αντιευθέτησης ε, διαφόρων και προσπαθήσαμε να τις προβάλλουμε ως μια στρατηγική πρωτοβουλία και να σας πω ότι στην πολιτική μας που είναι τρόφιμα και καταναλωτές Πρόκειται για, ένα, για μια στρατηγική πρωτοβουλία. Και αυτό καταδεικνύει τη σημασία του εγχειρήματο. Όπως είπε και ο Επίτροπος Ντάλι, θεωρούμε ότι προκειμένου να υπάρχει μια εύρυθμα λειτουργούσα αγορά, θα πρέπει να προσφέρουμε στον καταναλωτή τη δυνατότητα να έχει τέτοια δυνατότητα ε, με επίλυσης των διαφόρων. Είναι λοιπόν ε, σημαντικές οι εναλλακτικέ μέθοδοι, γιατί είναι φτηνές, γρήγορε γρήγορες ε, για τον καταναλωτή. Αλλά είναι και μια κατάσταση διπλού ωφέλους και για τις επιχειρήσεις, γιατί τους επιτρέπει να διατηρούν μια φήμη στην αγορά. Γιατί Φυσικά η αγορά βασίζεται σε δύο πυλώνες, και στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Αν λοιπόν δεν εμπιστεύονται οι καταναλωτές στις επιχειρήσεις, να λειτουργεί η αγορά. Όπως είπε και ο Επίτροπος, κατά την φάση της διαβούλευσης εξετάσαμε επειδή πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά προς επίλυση, για παράδειγμα πόσο μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση, μπορεί να καταστεί το ADR ένα πρώτο βήμα πριν τις ε, νόμιμες διαδικασίες, τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε στη φάση Α, της ε. Ε, διαβούλευσης πώς ε, θα διαμορφωθούν αυτά και φυσικά θα διαμορφωθούν και από τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας ευχαριστούμε Μάλκομ για την συνεχή σας υποστήριξη. Well, Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το πρώτο σχέδιο και ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και εσείς και η ομάδα σας. Αν υπομονούμε να δούμε και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Ε, να περάσουμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τέρι, ο οποίος θα ξεκινήσει την επόμενη, την κυρία Ευελίν Τέρι, η οποία θα ξεκινήσει την επόμενη παρουσίαση. Να διευκρινίσω απλά ότι θα τηρήσουμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα γιατί ο κανόνας που ακολουθώ στις ακροάσεις είναι να είμαστε αυστηροί με το χρόνο. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πέντε λεπτά στη διάθεσή τους. Θα είμαστε αυστηροί με το χρόνο ομιλίας. Θα βλέπετε μπροστά σας ε, πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας ακόμα. Να σας δώσω και το σφυράκι άμα θέλετε. Σας το δίνω, να για να υπενθυμίζετε στους συναδέλφους που μακρηγορούν ότι ενδεχομένως να χρειάζεται να είναι πιο λακωνική. Αυτά. Και σας δίνω το λόγο. Και εγώ θα πάω να κάτσω κάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι υπεύθυνη για το ρολόι, γιατί συνήθως είναι από την άλλη πλευρά και είμαι εγώ αυτή που περιορίζομαι. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα σε μια πολύ σημαντική τέτοια σύνοδο, σε μια πολύ σημαντική χρονική συγκυρία όπου λαμβάνονται πολύ σημαντικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά και σε ό,τι αφορά και τη συζήτηση προσανατολισμού που ακούσαμε πριν από λίγο. Ψηφίστηκαν τρεις ε, σημαντικές εκθέσεις σήμερα το πρωί στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα θα συζητήσουμε το ADR, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για του καταναλωτέ. Έχετε είναι πολύ ευρεία κλίμακα στα δικαιώματα του καταναλωτή στην Ευρώπη και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Αλλά αν τα δικαιώματα παραμένουν στη θεωρητική σφαίρα, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες ε, για το ADR. Το ακούσαμε αυτό πριν από λίγο και ακούσαμε επίσης ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα σε ό,τι αφορά το ADR. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Οι καταναλωτές ε, δεν απευθύνονται με τα προβλήματά τους σε ένα σώμα ADR. Άρα, ε, αν υπομονούμε να ακούσουμε τη σημερινή συζήτηση, ολοκληρώθηκε και η διαβούλευση χτες, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν και οι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, α, οι εμπλεκόμενοι φορεί και οι υπόλοιποι που συμμετέχετε στην παρούσα συνεδρίαση. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Σφαπ, Ευρωβουλευτή, μέλο τη Επιτροπής Εσωτερική Αγορά και Καταναλωτών και ο οποίο παρακολουθεί το θέμα αυτό εκ του συνεκής. Έχετε το λόγο λοιπόν να μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας για το ADR. Το πρώτο πάνελ θα επικεντρωθεί στα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ADR και το επόμενο πάνελ θα εξετάσει πιο πολύ τα μελλοντικά προβλήματα. Να ακούσουμε λοιπόν τη θέση σας. Thank you so much, uh, Professor Terin. Uh, so much for... Σας ευχαριστώ κυρία καθηγητά. Κυρία καθηγήτρια, συγγνώμη. Ε, οκ, okay, να είμαι λοιπόν σύντομος και σαφής. Πιστεύω και είναι βεβαίω και η ξεκάθαρη θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο ότι αυτό που έχει σημασία στην αγορά είναι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και κυρίω στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ένα σοβαρό μηχανισμό διευθέτηση των διαφορών είναι απολύτω κρίσιμος. Η πρόταση και η συζήτηση για την ελλακτική διευθέτηση διαφορών είναι πολύ σημαντική διότι πρόκειται για ένα μηχανισμό, ένα εργαλείο το οποίο είναι πολυμερό ενδιαφέρον δεν είναι γραφειοκρατικό, προσφέρει μεγάλη ευκαμψία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αποφεύγουν την επιβάρυνση μιας δικαστικής διαφοράς, που έχουμε δει και τις δυσκολίες με τις συλλογικές αγωγές στις ΗΠΑ, λειτουργεί και διαμεθοριακά, χωρίς να τίθεται θέμα εάν το ευρωπαϊκό επίπεδο έχει την αρμοδιότητα να νομοθετεί σε θέματα συλλογικών συστημάτων αποζημιώσεων, διότι βασίζονται αυτά συνήθως σε εθελοντικές συμφωνίες, προσφέρει ταχύες λύσεις και για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις, προσφέρει επίσης λύση χαμηλού κόστους και αυτά είναι πολύ θετικά. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε έναν αριθμό θεσμών, φορέων και κυρίως στον χώρο αρμοδιότητας του κυρίου Ντάλι, όπου μπορούμε να βασιστούμε. Στην δική μου εκλογική περιφέρεια, κοντά στο Στρασβούργο, στο ΚΕΛ δηλαδή, η, η οργάνωση εκεί έχει δείξει σημαντική δραστηριότητα και πώς μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές προσφέροντας ενημέρωση και δίνοντάς τους προσανατολισμό για να χρησιμοποιήσουν τους μηχανισμούς εναλλακτική διαθέτησης διαφορών. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξουν αυτά σημαντικό ρόλο, αλλά υπάρχουν ακόμα ορισμένε προκλήσεις. Πρώτον, πώ θα είναι διαφανή η διάρθρωση σε όλες τις χώρες μέλη. Γνωρίζουμε ότι τα συστήματα αυτά δεν ισχύουν ακόμη σε όλη την Ευρώπη. Αν θέλουμε όμως όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να μπορούν να υποφελούνται, πρέπει να διασφαλίσουμε μια πανευρωπαϊκή δομή. Δεύτερο, πώς μπορούμε να αποφύγουμε το one size fits all, ταυτόχρονα σε επιτρέποντα σε όλου του Ευρωπαίου καταναλωτέ να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα συστήματα. Και τρίτο και πολύ σημαντικό θα πρέπει να είναι η ουδετερότητα των μηχανισμών εναλλακτική διευθέτηση διαφορών. Διότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σύστημα που θα βάζει στο επίκεντρο των συζητήσεων το ενδιαφέρον, το συμφέρον του καταναλωτού και τίποτε άλλο. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλια που θα ακούσω σήμερα το απόγευμα, ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε τη δική μα θέση ακόμη πιο σαφή. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Η κυρία Τερίν, σα ευχαριστώ πολύ για την πραγματικά διαβιέστατη τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ και για το γεγονός ότι στεβαστήκατε απολύτως ε, τον χρόνο σας. Δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω το σφυράκι του Προέδρου. Η κυρία Χόιενς τώρα, Γενική Διευθύντρια της ΜΠΕΚ, που είναι η κεντρική οργάνωση της Ευρώπης, που θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα σχετικά θέματα, που είναι σημαντικά για τους καταναλωτές. Θα ακούσουμε με ενδιαφέρον γιατί κατά τη γνώμη σας οι μηχανισμοί της εναλλακτικής διαθέτησης διαφορών ακόμη δεν έχουν φτάσει σε πλήρη απόδοση υπέρ των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα δύο λεπτά του κυρίου Σουβά που δεν χρησιμοποίησε. Λοιπόν, τα έχω και ανάγκη. Τέλο πάντων, είμαστε σοβαροί. Ευχαριστώ που μα δίνετε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφή για το EDR και να δω, σας δώσω την άποψη των καταναλωτών. Πρέπει να σας πω από την πλευρά των καταναλωτών υπάρχουν ε, πάρα, πολλοί, ε, πάρα πολλές διαφορές και μη ικανοποιημένοι καταναλωτές και πολλοί έμποροι που δεν θέλουν να λύσουν τις διαφορές. Αυτή είναι η καθημερινή πραγματικότητα και αυτό είναι το ιστορικό και βάση αυτού του ιστορικού θα εξετάσουμε το θέμα. Οι οργανώσεις καταναλωτών βλέπουν το ADR σαν ένα πολύ καλό εργαλείο σε μια εργαλειοθήκη γενική όπου χρειάζονται οι καταναλωτές για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Έχει πάρα πολλά ωφέλη σε ε, σχέση με το παραδοσιακό δικαστικό σύστημα από τη στιγμή που εφαρμόζεται σωστά και χρησιμοποιεί όλα τα ωφέλη που μπορεί να δώσει ένα σύστημα ADR, εναλλακτικό σύστημα επιλύσεως διαφορών δηλαδή. Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι εναλλακτική λύση. Άρα πάντα υπάρχει η έννοια, εμπεριέχει την έννοια τη επιλογή. Δεν αντικαθιστά την προσφυγή στο δικαστήριο. Η προσφυγή στο δικαστήριο παρέχει μοναδικά χέγγια που δεν μπορεί να προσφέρει το εναλλακτικό σύστημα ε, επίλυση των διαφορών, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και αυτοί που διαφορούν την πολιτική πρέπει να επενδύσουν στο ADR, να γίνει όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται αυτό το εναλλακτικό με στη φύση των διαφορών, αλλά μην λησμονούν να επενδύουν στη βελτίωση των δικαστικών μηχανισμών αποζημιώσεω και διορθώσεω και επίλυση των διαφορών όπως είναι, για ε, είναι και τα μέτρα για τη συλλογική προσφυγή. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας παρατηρήσεις. Γιατί δεν χρησιμοποιείται πλήρω το ADR και δεν φτάνει στο πλήρω δυναμικό. Να τονίσω τρία πράγματα. Κάτι που ανέφερε και ο Επίτροπο Νταλή. Οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν καταρχά ότι υπάρχει αυτή η εναλλακτική μέθοδο επιλύση των διαφορών, το ADR. Δεν το επαναλάβω αυτό. Πέρα όμως ότι δεν το γνωρίζουν οι καταναλωτές, υπάρχει και σύγχυση που επικρατεί στους καταναλωτές, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά ε, σχήματα και μηχανισμοί, ονομασίες διαφορετικές, παρόμοιοι μηχανισμοί με παρόμοια ονομασία, οπότε ο κόσμος μπερδεύεται και χάνεται. Άρα να σχολιάσω κάτι, που είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Καμιά φορά οι υπηρεσίες ε, επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν τις, τα παράπονα είναι και, αυτοί, αυτές μπερδεύονται με τα συστήματα επίλυσης διαφορών και πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των σχημάτων EDR που είναι εξωτερικά και τα εσωτερικά που έχει κάθε εταιρεία. Ε, ενεργειακή εταιρεία. Η ZF Suez, ε, ε, η γαλλική για το φυσικό αέριο, έχει, έχει μεσολαβητή, λέγεται Mediator. Υπάρχει όμως μια μονάδα που εξετάζει παράπονα και στη Γαλλία το κοινοβούλιο δημιούργησε τον Mediator de l'Energie, διαμεσολαβητή φορέα δημόσιο για την ενέργεια. Άρα υπάρχει σύγχυση και πιστεύουμε ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να βοηθήσουν του καταναλωτέ να καταλάβουν καλύτερα, να υπάρχει σαφήνεια, να έχουν περισσότερε πληροφορίε για τα σχήματα EDR, ίσω να υπάρχει ένα πρότυπο, ένα σύστημα ενημέρωσης να τους δίνει, να του διαγραφεί, να του δείχνει τα συστήματα, να τα συγκρίνει, αυτή η παρουσίαση και να ξέρουν καλύτερα τι να κάνουν. Αλλά δεν χτυπάει με τον τηλέφωνο, ελπίζω όχι. Λοιπόν, όσον αφορά τι ονομασίε κλπ. Ε, άλλη παρατήρηση που σχετίζεται με τι πρώτε. Οι κατανοητέ δεν γνωρίζουν διότι οι έμποροι το χρησιμοποιούν. Αν οι έμποροι χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά και πρότειναν τα σχήματα EDR, τότε οι κατανοητέ θα τα γνώριζαν περισσότερο. Όπω είπε ο κύριο Νταλή, μόνο 40% των εμπόρων, των εμπορευμένων το γνωρίζουν και αν το γνωρίζει το σύστημα το χρησιμοποιούν. Γιατί το χρησιμοποιούν για να είμαι και κάπως προκλητική. Δεν το χρησιμοποιούν το σύστημα διότι δεν έχουν κίνητρο να το χρησιμοποιήσουν. Διότι αν υπήρχε ε, κάποια απειλή, αν ξέρανε ότι ο καταναλωτής, μάλλον ήξεραν, υπήρχε ένα δέλεαρ και ξέρανε ότι δεν... Ε, Μάλλον υπήρχε απειλή. Ο καταναλωτή θα πάει στο δικαστήριο. Αν δεν του προταθεί το ADR, τότε θα το πρότειναν το ADR. Μετά υπάρχει και έλλειψη συμμόρφωση από τι επιχειρήσει. Υπάρχουν σχήματα ADR τα οποία είναι δεσμευτικά για του εμπορευόμενου. Υπάρχουν σχήματα ADR που δεν είναι δεσμευτικά. Η απόφαση δεν είναι δεσμευτική για τον εμπορευόμενο. Αυτό εξαρτάται τότε για, στην καλή βούληση του εμπορευόμενου. Υπάρχουν βέβαια επιχειρήσει που συμμορφώνονται πλήρω με την απόφαση των διαφόρων μηχανισμών ADR, αλλά υπάρχουν άλλε εταιρείε που δεν τι νοιάζει καθόλου. Πώ τα βλέπει τώρα ο καταναλωτή. Εδώ είναι κολυσιεργή αυτό. Δηλαδή, περνά από όλη τη διαδικασία από το σύστημα και στο τέλο πάλι έχεις χάσει. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνοι που διαμορφώνουν την πολιτική θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα όπου στο μέτρο του δυνατού η απόφαση που λαμβάνει ο μηχανισμός δεσμεύει τον εμπορευόμενο. Κατακλείδη να πω ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όπως ο κύριος Εφαλβάη όσον αφορά την αυτονομία, αυτόνομο έλεγχο της αγοράς όσον αφορά τη θέση των διαφορών. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία στους μηχανισμούς ADR αλλά για να λειτουργεί το σύστημα, να έχει την έγκριση, την εξουσία να μπορεί να θεωρηθεί ω τέτοιο, πρέπει να πληρούνται κάποιε προποθέσει και να γίνονται σεβαστέ, ούτω ώστε πραγματικά αυτό ο μηχανισμό να δίνει στον καταναλωτή ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο και ότι κάπου θα καταλήξει. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χόιεντ. ευχαριστώ που επισημάνατε και το σημαντικό πρόβλημα αυτό της ε, ευαισθητοποίησης και σε ό,τι αφορά τη συμπληρωματικότητα των ε, συστημάτων ADR. Είναι πολύ σημαντικός ο μηχανισμός. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκρέκο, ο οποίος είναι επίσης ευρωβουλευτές, μέλος της Επιτροπής ε, ΙΜΚΟ και ήταν και εισηγητής της σημαντικής έκθεσης για την ενιαία αγορά για τους καταναλωτές, όπου τονίσατε την ε, ευθύνη και το ρόλο των καταναλωτών και των πολιτών σε μια ενιαία αγορά. Αναφερθήκατε και εσείς στο θέμα του ADR και της ε, περιορισμένης ε, ευαισθητοποίησης του κοινού. Να ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις σας για τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ADR. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον Επίτροπο και τον Υπουργό ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, σε όλη την Ευρώπη δεν καταλαβαίνουν ε, απόλυτα ούτε γνωρίζουν τα συστήματα, τα ε, σχήματα ADR. Λίγοι μόνοι πολίτες ξέρουν πώς μπορούν να αποτανθούν σε ένα τέτοιο σώμα ADR. Κάποιοι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει τέτοια μορφή ε, υποβολή ενστάσεων. Είναι σημαντικό λοιπόν η, τα σχήματα αυτά διευθέτησης διαφορών που δεν λειτουργούν ακόμα σωστά για να δίνουν ε, στους Ευρωπαίους πολίτες ε, έναν γρήγορο και αποτελεσματικό εξοδικαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Είναι κατακαιρματισμένο λοιπόν το περιβάλλον σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια λόγω έλλειψη ε, πληροφοριών. Είναι κατακαιρματισμένο το σύστημα, δεν υπάρχουν νομοθετικέ πρωτοβουλίε και δεν υπάρχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Όλα αυτά λοιπόν ε, παρεμποδίζουν τους ε, καταναλωτές από τη χρήση των συστημάτων ADR. Θα έπρεπε να υπάρχει πιο μεγάλη ασφάλεια, πιο μεγάλη αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά καταναλωτέ που αντιμετωπίζουν διαρκώ δυσκολίε σε διασυνοριακές ε, περιπτώσεις. Παρόλο που δεν απευθυνόμαστε σήμερα σε θέματα συλλογικών αγωγών, θεωρώ ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και ένας μηχανισμός συλλογικής αγωγής για να συμπληρωθούν οι αναλεκτικές μέθοδοι ε, διευθέτηση διαφορών. θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα συλλογικής αγωγής ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως πρότεινε και η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του περσινού έτους. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις εφιστάμενες δομές, ιδιαίτερα τα δίκτυα ECC, και να φροντίσουμε να έχουν τους απαραίτητους πόρους, την απαραίτητα χρηματοδότηση προκειμένου να λειτουργούν αποτελεσματικά και προκειμένου η στρατηγική ενημέρωση να εξηγήσει τις λεπτομέρειες του συστήματος στους πολίτες προκειμένου εν, ενδεχομένως να ενσωματώσει και τα συστήματα ενημέρωσης περί ιστορικής αγοράς στο τελικό πακέτο ADR. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσον ένα αναθεωρημένο σύστημα ADR θα περιλάβει και τις, ε, τις ε, συναλλαγές μεταξύ, μεταξύ επιχειρήσεων ή μόνο τις ε, συναλλαγές καταναλωτή με επιχειρήσεις. Ζήτησα να εξεταστεί πώς οι πολίτες και οι μικρόμεσαίες επιχειρήσεις και οι καταναλωτές ασκούν τα δικαιώματά τους και να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια στοχευμένη μια στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι διασυνοριακές συναλλαγέ και την κυκλοφορία των αποτελεσματικών πληροφοριών, την ενημέρωση. Καταλαβαίνω, κυρία Πρόεδρε, ότι το θέμα αυτό είναι περίπλοκο και πολύ σύνθετο ακόμα και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό οποιοδήποτε σύστημα που θα περάσει θα πρέπει να περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλεία κατά των καταχρήσεων και κατά ανεύθυνων συμπεριφορών μετά από ακροάσεις, εκθέσεις, σεμινάρια. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει. Καλό λοιπόν τον Επίτροπο Ντάλι και την υπηρεσία του να μην καθυστερήσει στην ε, ολοκλήρωση του πακέτου αυτού, να κάνει μέχρι το τέλος του 2011 μία συγκεκριμένη πρόταση για το ADR και για ένα μηχανισμό συλλογικής αγωγής. Θα πρέπει να δυσφαλιστεί ότι το σύστημα το οποίο τελικά θα περάσει θα είναι βιώσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την έκκλησή σας και για την επισκόπηση που μας δώσατε των σημερινών προβλημάτων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φρίζο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις ο οποίος είναι διαμεσολαβητής στον ασφαλιστικό, στον ασφαλιστικό κλάδο και μέλος του FINET. Όπως θα ξέρετε, πρόκειται για ένα σώμα, μια ένωση α, υπηρεσιών ADR. Ανυπομονούμε να ακούσουμε λοιπόν τις δικές σας προσωπικές απόψεις και εμπειρίες και να μας πείτε πώς λειτουργεί η Φιλανδία. Ίσως να μας δώσετε και κάποια παραδείγματα επιτυχίας στην Φιλανδία δράτω με της ευκαιρίας που μου δίδεται για να εκφραστώ γαλλιστή για μια φορά σε αυτό το βήμα. Ε, Είναι πιο απλό για μένα για να εκφράσω την εμπειρία που έχω ως διαμεσολαβητής του ασφαλιστικού τομέα στη Γαλλία εντός του δικτύου Fitnet. Στο σύντομο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μου θα υπενθυμίσω εν συντομία κάποια ιστορικά στοιχεία, πώς λειτουργούμε, και μετά θα δώσω και κάποια παραδείγματα. Καταρχάς, γιατί Φιλνέτ, η ανάγκη που υπάρχει στον τομέα το χρηματοστατικό για να δημιουργηθεί ισορροπία εκ νέου μετά το άνοιγμα και τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς επιβάλλεται κάτι πολύ γρήγορα μάλιστα. Ήταν πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να μπορούν να προσφύγουν σε ένα μηχανισμό ο οποίος θα τους επέτρεπε να έχουν ταχεία πρόσβαση σε μια κάποια μορφή δικαιοσύνης. Ποια είναι η κεντρική ιδέα, η γενική ιδέα. Λοιπόν, θέλαμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, το οποίο δίκτυο θα επέτρεπε να ρυθμιστεί χωρίς να χρειάζεται προσφυγή σε δικαστικές διαδικασίες όταν υπάρχουν δαπάνη, ε, ε, μηχανισμοί, ένας μηχανισμός λέγω που θα διευθετεί τις διαφορές τις οικονομικές, τις διασυνοριακές. Το FINET απαρτίζεται από διάφορα συστήματα ADR που έχουν δημιουργηθεί στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και όπου ήδη έχουν επιφορτιστεί με την επίλυση των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και των παρόχων χρηματοσυντικών υπηρεσιών, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και του χρηματοστητικού τομέα της αγοράς. Οι μηχανισμοί ADR εντός της του FinET συνεργάζονται για να διευκολύνουν την πρόσβαση του καταναλωτή και να μπορούν σε περίπτωση διαφοράς οι καταναλωτές να απευθύνονται στο σύστημα το εγκύτερο το οποίο θα έρθει σε επαφή ε, με το ομόλογο σύστημα στη συγκεκριμένη χώρα ούτω ώστε να ε, ρυθμιστεί το θέμα το ταχύτερο δυνατόν. Η δημιουργία λοιπόν του δικτύου γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τους υφιστάμενους μηχανισμούς. Η ιδέα δεν ήταν να αρμονιστούν τα διάφορα συστήματα, αλλά να ενωθούν εντός ενός δικτύου συνεργασίας άνευ ε, ρυθμίσεων της ενώσεως. Και τέλος, διευκόλυνση στο μέγιστο βαθμό της συγκεκριμένης λύσεως επιλύσεως των διαφορών, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία εντός του δικτύου. Το FINET e δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2001 μετά από μια περίοδο άτυπων συνεδριάσεων ε, και λειτουργίας των ανεπισήμων συστημάτων. Σήμερα 50 μέλη από 22 χώρες συμμετέχουν στο δίκτυο και υπάρχει πρωτόκολλο συμφωνίας που αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασυνοριακών Προσφυγών στον τομέα των χρηματοστατικών υπηρεσιών που το MOM. Το... Α, είναι το υπόμνημα συνεννόηση αυτό το πρωτόκολλο. Το μνημόνιο συνεννόηση. Αναλύει τη διαδικασία, το μνημόνιο, δηλαδή πώ χρησιμοποιείται το εγκύτερο σύστημα EDR, το πιο κοντά στον καταναλωτή, που με τη σειρά του αυτό το σύστημα θα απευθυνθεί το αρμόδιο σύστημα για να αντιμετωπιστεί η υπόθεση ε, που αφορά και τον πάροχο τη υπηρεσία. Λοιπόν, ε, χρησιμοποιείται η γλώσσα τη συμβάσεω, η αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην αλλαγή και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ADR αλλά επίσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι το σημαντικό σημείο που θέλω να επιμείνω. Είναι η ποιότητα των παρεμβάσεων. Ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει ύψιστη ποιότητα επεξεργασίας των διαφορών για να κερδίσουμε και να διονύσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτού σε ένα τέτοιο δίκτυο ADR. Βεβαίως υπάρχουν οι ίδιες οι αρχές της συστάσεως του 98 και του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελήφθησαν υπόψη όπως και στην οδηγία του 2008 για τις εμπορικές συναλλαγές, στη σχετική οδηγία έλήφθησαν υπόψη. Βασικές αρχές γίναν σεβαστές. Ακολουθούν οι φορείς για την επίλυση των διαφορών αυτές τις αρχές. Και είναι κάτι που χρησιμοποιούν τα ADR. E Συνεχώς σέβονται τις αρχές αυτές. Είναι προπόθεση άλλωστε για την κοινοποίηση του συστήματο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τι κυβερνήσει των κρατών μελών. Και αυτή η κοινοποίηση επιτρέπει το ADR το συγκεκριμένο να ενταχθεί στο δίκτυο FINET. Αυτές οι αρχές είναι πυλώνε σοφίας αν θέλετε. Ανεξαρτησία του δημοσιολογητή απαιτείται. Διαφάνεια των αστηριοτήτων. Αποτελεσματικότητα. σεβασμό τη νομιμότητα, ισότητα, Ελευθερία για επιλογή της διαμεσολάβησης αντί της δικαστικής παρέμβασης, προσφυγή στην ισότιμη αντιμετώπιση, σεβασμός της αντίφασης, της αντιπαράθεσης, σεβασμός του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στοιχείων και δωρεάν ή ιονή δωρεάν παροχή των υπηρεσιών στον καταναλωτή. Ελεύθερη πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα διαμεσολάβησης. Πετύχαμε, κατά την άποψή μου ναι, ο αριθμός τον ADR εντό του FINET, το δείχνει αυτό, ε, ήταν λιγότερο από 1500, 1500 υποθέσεις αντιμετωπίστων 2.000, σήμερα εξετάσαμε 7.000 στο FINET υποθέσεις με πάνω από 1.500 θέματα μέσω όρο το έτος τα τελευταία χρόνια. Αυτό το δίκτυο δεν είναι πάντα γνωστό, αρκετά γνωστό θα έλεγα. Είναι το βασικό συμπεράσμα της εκθέσεως τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολόγησε το FINET έκθεση που ετοιμάστηκε το Φεβρουάριο του 2009 και τα συμπεράσματα ποια ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αντιτικοποιήσει την πρόθεση του δικτύου και να διοργανώνει ταυτόχρονα τη, διοργάνωση, τη διεύρυνσή του, να συμπεριλαμβάνει περισσότερα μέλη. Λοιπόν, και σε εθνικό επίπεδο γίνεται η πρόθεση του ΦΙΝΕΤ και δημιουργείται επαφή με, τα το διεθνέ Δίκτυο Info που συμπεριλαμβάνει του χρηματοστικού δημοσιολαβητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είμαι μέλο τη Διευθύνουσα Επιτροπής του Δικτύου με το φίλο μου, το, διαμεσολαβητή, τον οικονομικό, το χρηματοστικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Το FINET έχει στο σελίδα που συμπεριλαμβάνει τη βάση δεδομένων σε πολλέ γλώσσε, μόνε πληροφορίε που αφορούν τα συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τέλος η έκταση αστηριοτήτων του δικτύου στην ίδια ιστοσελίδα σελίδα φαίνεται ε, νομίζω ότι δεν μπορώ να παραθέσω τα παραδείγματα που ήθελα διότι μου τελείωσε ο χρόνος. Μπορείτε να δείτε τα παραδείγματα τα συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα που σας ανέφερα στην παρεμβασία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φριζόν. Ευχαριστώ που λίγο πολύ τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα. Ε, μας εξηγήσατε το λόγο ύπαρξης του ΦΙΝΕΤ, πώς λειτουργεί, Συγκεκριμένα στοιχεία μας δώσατε επίσης όσον αφορά τη λειτουργία του, του συστήματος FinNet. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Diana Wallis, που είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που γνωρίζει το ADR πολύ καλά, το παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ, άρα ενδιαφερόμαστε πολύ να ακούσουμε ποιε είναι οι απόψει σα όσον αφορά το σύστημα αυτό, το εναλλακτικό σύστημα επιλύση των διαφορών, η ADR. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, μου σε ευχαριστώ και τον Επίτροπο που αναζωογόνησε, ας πούμε έτσι, το θέμα, διότι προπαρασκευαζόμενοι για τη σημερινή διάσκεψη ξανακοίταξα τα αρχεία μου και είχα κάνει σχετική έκθεση το 2001. Θα ήθελα να είχαμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε προχωρήσει, αλλά τέλος πάντων εύχομαι σε όλους κουράγιο για την περαιτέρω προσπάθεια. Η αξία της εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών μου φάνηκε καθαρά από κάποιον που μου έγραψε και στην εκλογική μου περιφέρεια δηλαδή και μου είπε είμαι Ιταλός συνταξιούχος είμαι σταξιούχος μάλλον στην Ιταλία, δεν βγάζω άκρη. Βάλαμε το σύστημα στο, βάλαμε την ερώτηση μάλλον στο Solvit και είδαμε ότι είχε προσπαθήσει δυόμιση χρόνια να ε, λύσει το πρόβλημά του, το Solvit το έλυσε αμέσως. Και τώρα ε, το πρόσωπο αυτό είναι πλέον φανατικός οπαδός και του Solvit και του ADR. Πώς μπορούμε τώρα να φέρουμε τα συστήματα αυτά και σε άλλους τομείς όπως αυτούς που συζητούμε τώρα και ε, στο έγγραφο της διαβουλεύσεως υπάρχουν ακόμα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το πρώτο και μεγαλύτερο νομίζω είναι πραγματικά η ευαισθητοποίηση. Ο κόσμος γνωρίζει που βρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο, γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί για να ζητήσει αποζημίωση. Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο φάσμα συστημάτων εναλλακτική διευθέτηση διαφορών που από σε ένα επίπεδο είναι καλά, αλλά σε ό,τι αφορά αν γνωρίζει ο κόσμος πού πρέπει να απευθυνθεί, δεν είναι καλά. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κάποια διέξοδο, κάποιο δρόμο που να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα υπέρ των πολιτών. <clears throat> Θεωρώ ότι μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουμε. Θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε έναν οδικό χάρτη συνεκτικό που να διασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτέ μπορούν να φτάσουν στο σύστημα εναλλακτική διευθέτηση διαφορών που θα αποδώσει, που θα του προσφέρει αποτελέσματα. Είχαμε τον κώδικα δεοντολογίας, είχαμε και το μνημόνιο Συμφωνία που έχουν περάσει από τα διάφορα γραφεία ε, στο παρελθόν. Δεν φαίνεται όμως να, να μπόρεσαν να μας οδηγήσουν οι μηχανισμοί αυτοί εκεί όπου θέλαμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι το πλέον στιβαρό, αν μπορώ να το πω έτσι, για το μέλλον. Και νομίζω Οπότε έχει δίκιο όταν λέει ότι χρειαζόμαστε κάτι που θα εμπλέξει περισσότερο τις επιχειρήσεις. Ένα καλό σύστημα εναλλακτική διευθέτησης διαφορών θα πρέπει να είναι, να ενταχθεί μέσα στην συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Άλλο βέβαια είναι η εξυπηρέτηση των πελατών και άλλο είναι το ADR. Πρέπει όμως να είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι χρήσιμο και για αυτές. Εν τέλει θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί, να μελετήσει και την έκθεση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κρίση της ασφαλιστικής εταιρείας Equitable Life. Το ίδιο σενάριο δεν γνώριζαν οι άνθρωποι τότε αν έπρεπε να πάνε στους εθνικούς διαμεσολαβητές σε μία χώρα ή σε άλλη χώρα. Πήγαιναν από, τον Άννα στον Καϊάφα. Τελικά μπορέσαμε κάποια πράγματα να διευθετήσουμε, αλλά είτε δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, υπάρχει και ένα βέβαια πρόβλημα πόρων για το FinNet. Η εναλλακτική διευθέτηση διαφορών δεν είναι απονομή δικαιοσύνη με χαμηλό κόστος θα πρέπει για να λειτουργήσει σωστά να έχει και σωστή επαρκή χρηματοδότηση. Το σενάριο της Equitable Life μας έδειξε καθαρά ότι εάν θέλουμε να έχουμε πραγματική πρόσβαση σε αποζημιώσεις, σε δικαιοσύνη, σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, δεν χρειαζόμαστε μόνο μηχανισμούς εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι μάλιστα και συμπληρωματική σε ένα καλό σύστημα συλλογικών αποζημιώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν αλληλοαποκλείονται, είναι αλληλοσυμπληρώμενα τα συστήματα αυτά. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε για το ότι παρακολουθείτε το σύστημα αυτό ADR και για τις δράσεις που έχετε αναλάβει. Υπογραμμίσατε ότι υπάρχουν όντως, μάλλον υπογραμμίσατε πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα. Για παράδειγμα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για να βρουν το κατάλληλο όργανο ADR στο οποίο πρέπει να αποτανθούν. Και αυτό ασφαλώς αποτελεί και ένα, μία από τις προκλήσεις αναφορικά με το ADR. Επίσης, ε, υπογραμμίσατε την πρόκληση του να εμπλεχθούν και οι εταιρείε και τα πλέον εκτίματα που θα σημαίνει αυτό για τις εταιρείε. Τελευταίος ομιλητής, τελευταία μάλλον ομιλήτρια, πρώτη δώσουμε το λόγο στην αίθουσα, η κυρία Πόμπη, από πλευράς των επιχειρήσεων, αντιπρόεδρος της ε, Ιταλικής Ένωσης ε, του Ιταλικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Επιμελητηρίου, να ακούσουμε τις απόψεις σας, γιατί στην παρούσα φάση μόνο το 9% των λιανικών επιχειρήσεων έχουν χρησιμοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ADR. Γιατί λοιπόν οι επιχειρήσεις ε, διστάζουν να χρησιμοποιήσουν το ADR. Καλησπέρα ζητώ συγγνώμη γιατί θα μιλήσω Ιταλικά, αλλά υπόσχομαι ότι θα τηρήσω το χρόνο που μου διαθέσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας μεταβιβάσω την Ιταλική εμπειρία και των Ιταλικών εμπορικών επιμελητηρίων. Τα Ιταλικά ε, ε, εμπορικά επιμελητήρια είναι δημόσια πρόσωπα και παίζουν ρόλο διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων και των καταναλωτών ένα ρόλο τρίτου μέρους και ανεξαρτησίας και όσον αφορά ε, και την, ε, το ρόλο του που παίζουν σαν διαμεσολαβητής. Είναι ένα δίκτυο τα εμπορικά επιμελητήρια στην Ιταλία, ένα δίκτυο υπηρεσιών και λειτουργούν πάνω απ' όλα στην εθνική επικράτεια με κανόνες ομοιογενείς, με τέλη ομοιογενή και συμπεριφορά και ε, ομοιόμορφη. Είναι ιδιαίτερη κατά στην Ιταλία με ένα νόμο που εγκρίθηκε τον περασμένο Μάρτιο και επί τη βάση της οδηγίας της κοινοτικής η οποία επανειλημμένα αναφέρθηκε αυτή του 2008, η διαμεσολάβηση γίνεται υποχρεωτική και γίνεται υποχρεωτική ε, επί κάποιων θεμάτων όπως είναι διαδοχή, κληρονομιά, μίσθωση, ασφαλιστικά συμβόλαια, όλα αυτά που εμπλέκουν και τις εταιρείε και τους καταναλωτές. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πριν ξεκινήσει η διαμεσολάβηση, πριν πάει κανεί στο δικαστή, θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία μεσολάβησης. Άρα θα πρέπει να γίνει μια τέτοια απόπειρα και πρέπει να γίνει μέσω των φορέων εκείνων που είναι γεγραμμένοι σε ένα μητρό που είναι στο Υπουργείο, ε, καταχωρημένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε αυτό το ε, πλαίσιο λειτουργούν τα Ιταλικά επιμελητήρια. Είναι 105. Από τα 105 πάνω από 60 είναι γεγραμμένα στο Μητρό που σας ανέφερα. Και τα επιμελητήρια είναι σημαντική εμπειρία όσον αφορά τη διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων καταναλωτών. Τα τελευταία χρόνια υπήρχαν φορεί ε, που διαχειρίστηκαν με επίμαχο τρόπο. Ε, Είχαμε πάρα πολλέ διαφορέ. 80.000 στα 10 χρόνια και με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό που αξίζει τον κόπο να υπογραμμιστεί είναι ότι μία διαφορά από τις δύο επιλύεται σε λιγότερο από δύο μήνες. Και όχι μόνο για μικρές διαφορές, που αφορούν τους καταναλωτές και μιλάω και για τις διαφορές που αφορούν τις επιχειρήσεις. Και όχι μόνο αυτό όμως, δεν είναι μόνο υποχρεωτική αυτή η μεσολάβηση, αλλά γίνεται, είναι δυνητική η χρήση αυτή που συμπεριλαμβάνεται. Δηλαδή τα δύο μέρη δέχονται να μπουν ε, στη μεσολα... διαμεσολάβηση, μέσω της ρίζας διαμεσολάβησης. Ποια μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της διαμεσολάβησης. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά λοιπόν. Σίγουρα η ταχύτητα, η διαμεσολάβηση στην Ιταλία διαρκεί κατά ε, μέσο όρο 60 μέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία Ιταλικά. Ε, ενώ αν, σε αστικό δίκαιο πάει, πάμε στις 1200 μέρες στο δικαστήριο, το αστικό. Και ε, είναι μειωμένο το κόστος στη διαμεσολάβηση, στη διευθέτηση των διαφορών. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, είναι σημαντικό κίνητρο τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε στην Ιταλία, για μια εταιρεία το κόστος να πάει στη δικαιοσύνη σε ένα χρόνο είναι πάνω από 3.800 ευρώ. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο όσον αφορά. Ε, εγγυάται την αμερόληπτη προσέγγιση για τα μέρη. Είναι ευέλικτη διαδικασία όπου τα μέρη χειρίζονται τα ίδια τη διαμεσολάβηση και συνοδεύονται, επικουρούνται από ένα διαμεσολαβητή που προσπαθεί να βρει λύσεις σε αυτή τη διαφορά. Και αυτό βοηθά ε, τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Ε, περισσότερο το να διατηρηθούν οι σχέσεις παρά να διακοπούν. Αυτό, σε αυτό βοηθάει η διαμεσολάβηση. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι τη συμφιλίωση της λύσης των διαφορών online που θα βοηθούσε κάτι τέτοιο να διαδοθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην Ιταλία τα εμπορικά επιμελητήρια ε, πειραματίζονται ε, σε αυτό το τομέα τη διαμεσολάβηση επίλυση διαφορών online. Στην Ιταλία, εντό πέντε ημερών, εντός, εντός πέντε ημερών θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό τη υποχρεωτική επίλυση των διαφορών, τη διαμεσολάβηση. Και αυτό έγινε δυνατόν από σημαντική τοποθέτηση όχι μόνο των εμπορικών επιμελητηρίων, αλλά και από πλευρά των ενώσεων που εκπροσωπούν διάφορου επαγγελματικού κύκλου και κατηγορίε εκλήθη ε, η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτή τη μεταρρύθμιση και να προχωρήσει στο δρόμο αυτό του υποχρεωτικού χαρακτήρα της μεσολάβησης και αυτό με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών επιλύσεως των διαφορών. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, στόχος μάλλον. Όχι μόνο να χρησιμοποιείται περισσότερο αυτή η συνδιαλλαγή και συμφιλίωση, αλλά να δημιουργηθεί και ένα αποτέλεσμα πολιτισμικό, να διαδοθεί το εργαλείο αν είναι υποχρεωτικό θα χρησιμοποιείται από όλου το μέτρο και έτσι όλοι θα το μάθουν το μέσο αυτό, θα θέλουν να το χρησιμοποιούν εκ νέου και για άλλες περιπτώσεις διαφορών. Αυτό σημαίνει από τις 90.000 διαφορές ε, θα πάμε στις 600.000 διαφορές. Τόσο, αυτή θα είναι η συνέπεια για τον επόμενο χρόνο, από 90-600.000 διαθετήσεις. Λοιπόν, γίνεται αυτή η προσπάθεια οι περισσότερες επιλύσεις, διευθετήσεις αφορούν τις τηλεπικοινωνίες στην Ιταλία. Στην Ιταλία διαμεσολαβήσεις όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και είναι και το θέμα αυτό, διάδοση και γνωστοποίηση του μέσου μέσω του υποχρεωτικού χαρακτήρα. Οι ρήτρε που μπαίνουν σε συμβάσεις το αναφέρουν αυτό. Διότι και αυτή η ρήτρα επιτρέπει την γνωστοποίηση του μέσου και μετά έχουμε τι κανόνε. Οι κανόνε είναι σημαντικοί. Κανόνε που δίνουν κίνητρα για τη χρήση. Φορολογικοί κανόνε, οικονομικοί κανόνε μάλλον, και οι κανόνε που καθιστούν δεσμευτική εκτελέση με την απόφαση δημοσιοληπτή. Όπω, παραδείγματο χάρη, ε, το θέμα τη έγκριση και επικύρωση των πρακτικών τη ε, διαμεσολάβηση, τη επίλυση αυτή των διαφορών. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή μαρτυρία για την κατάσταση που επικρατεί στην Ιταλία και τι εμπειρίε που θα καταστούσαν το ADR υποχρεωτικό. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις απόψεις που μας παρουσίασαν. Και τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε και άλλες μαρτυρίες, εμπειρίες προσωπικές από εκπροσώπους ε, ενώσεων καταναλωτών ε, του Κοινοβουλίου κάτι τελευταίο πρωτού ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Χάρμπαρ για να ε, προεδρεύσει κατά την φάση των συζητήσεων θα επικεντρωθούμε τώρα στην τρέχουσα κατάσταση και όλες οι ερωτήσεις για το πώς θα εξελιχθεί μελλοντικά το σύστημα ίσως καλύτερα να τεθούν αργότερα στο επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Εβελίν για την συντονισμό στο πρώτο τμήμα. Θα πρέπει να συντονίσω εγώ τώρα τον γύρο των ερωταπαντήσεων μιας και γνωρίσω και τους ε, ομιλητέ, αλλά θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Τζον Ντάλι και τον Υπουργό την παρατεστόρη, συγγνώμη, ε, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν, να πάνε σε μια σημαντική συνεδρίαση, να προασπιστούν τον προπολογισμό τους. Καταλαβαίνουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία και για τη σημερινή ε, συνάντηση. Μιας και είναι εδώ όμω ο κύριο Σεφαλβέη, θα του δώσω την ευκαιρία να απαντήσει σε ενδεχόμενα σχόλια. Έχετε το λόγο, συνάδελφοι να ρωτήσω αν κάποιοι συνάδελφοι ευρωβουλευτές θα ήθελαν να ξεκινήσουν τη συζήτηση με περαιτέρω σχόλια. Αλλά επίσης, αν θα ήθελαν και κάποιοι από το κοινό να σηκώσουν το χέρι τους, βλέπω κάποιους που σηκώνουν ήδη το χέρι τους, θα δώσω το λόγο καταρχάς ε, στους ευρωβουλευτές και δυστυχώ επειδή δεν ξέρω τα ονόματά σας και ακριβώ που κάθεστε θα σας ε, καλώ με τον αριθμό του έδρανού σας. Ξέρω ποιοι είσαστε λίγο πολύ, αλλά πρώτα να δώσω το λόγο στους βουλευτές. Και θα ήθελα οι ερωτήσεις, ε, αν γίνεται, να μην ξεπερνούν τα δύο λεπτά. εντεκτικό αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Τζοβάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από αυτό το πρώτο τμήμα, λέει και ο Ζουβέ, βλέπω ότι όλοι θέλουν να προστατεύσουμε καλύτερα τον καταναλωτή. Συμφωνούμε. Αυτό είναι κάτι καλό ήδη. Υπάρχουν ε, μηχανισμοί σε πολλά κράτη-μέλη, πάρα πολύ διαφορετικοί μηχανισμοί. Και τρίτον, παρατηρώ ότι ουσιαστικά πρέπει στο μέλλον, ακόμα και ξέρω ότι θα συζητήσουμε το μέλλον αργότερα, στο μέλλον λέω, θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει να εφαρμόσουμε διαδικασίε που αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση. Και κάτι που είναι και πιο περίπλοκο μετά, όταν μιλάμε για συλλογική προσφυγή, χρησιμοποιήθηκε αυτή ε, η διατύπωση, ε, κάποιοι εξέφρασαν και φόβους λοιπόν. Υπάρχουν πολλά είδη ε, αδράσεις και χρωστάμε στους συμπολίτε μας τη διαφάνεια όσον αφορά του ορισμούς. Και αληθεύει ότι αυτά που παρουσιάστηκαν από τους διάφορους παρεμβαίνοντες και από τους συναδέλφους τους βουλευτές είναι ότι όλη η ιστορία του, η ιστορία του Κοινοβουλίου ε, είναι μακρά όσον αφορά το θέμα αυτό και έχουν δοθεί πάρα πολλοί ορισμοί. Η Επιτροπή Ιστορικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτού πρέπει να βρει μια λύση όπου όλοι θα κερδίσουν. Να μην υπάρξει γενική πτώχευση αν θέλετε, όπως οι συλλογικές προσφύγες σε χώρες που γνωρίζουμε όπου έχουν βρει κάποια λύση μεταρρυθμίζοντας τα συστήματα που εφαρμόζανε όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. ορίμασαν τα πράγματα. Πρέπει να προσαρμοστεί δεόντως η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έγιναν κάποια εθνικά πειράματα. Τελείωσε αυτή η εποχή και πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ευχαριστώ τους διάφορους ομιλητές που αναφέρθηκαν στις διάφορες δοκιμές, την εμπειρία τους και στις εμπειρίες που έχουν, γίνει, ε, που έχουν οι διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και Ζουβέν. Η κυρία Ράπτη νομίζω είναι η επόμενη. Έχετε το λόγο κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας για τα πολύτιμα στοιχεία που μας έδωσαν. Παίρνω αφορμή από κάτι που είπε η κυρία Πομπέη. Ε, ζήτησε συγνώμη γιατί θα μιλούσε στην, ελληνική, στην Ιταλική γλώσσα. Ε, εκτιμώ την ευγένειά της, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει συγνώμη γιατί ζούμε σε μια πολυγλωσσική Ευρώπη. Έχουμε εξαιρετικούς μεταφραστές που μας βοηθούν καταπληκτικά στο έργο μας και η γλώσσα του καθενός μας είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Λέγοντας όλο αυτό, θέλω να επισημάνω, όπως είπαν και κάποιοι από τους ομιλητές, τη σημασία που έχει η γλώσσα στην επίλυση των διαφορών, ιδιαίτερα των διασυνοριακών. Και κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, διότι σε προηγούμενες συνεδριάσεις μου έχετε δώσει χρόνο μιλίας για όλη την τετραετία νομίζω, είναι κάτι που ξέρουμε εγώ και ο Πρόεδρος, ε, θέλω να πω ότι το θέμα του δικαιώματος στις συλλογικέ προσφυγές και το θέμα της ενημέρωσης για μένα είναι κομβικότατα σημεία για να προχωρήσουμε προς όφελος του καταναλωτή. Κλείνοντας δε, να πω ότι εκφράζομαι απολύτως από την εισήγηση που έκανε ο συνάδελφός μου κύριο Γκρέχ, κύριος Γκρέχ και ότι εκτίμησα εξαιρετικά την εισήγηση της κυρίας Βόλης. Ευχαριστώ. Well, thank you very much, uh, Rapti. Σας ευχαριστούμε κυρία Ράπτη και θα δώσω το λόγο να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας και στα ε, μέλη του Κοινοβουλίου να μας μιλήσει ο κύριος Φριζόν και να μας πει ε, ποιες είναι οι εμπειρίες του από ένα διευρωπαϊκό τέτοιο σύστημα. Να δω μόνο μήπως θέλουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι να πάρουν το λόγο πρώτα. Καταρχάς οι βουλευτές. Δύο κύριοι εκεί πίσω. Ο κύριος τα 153 και στο 196 που κάθεται από πίσω του. Και πολύ λυπάμαι που σας αποκαλώ με αριθμούς, αλλά αν θα θέλετε να συστηθείτε και από πού είσαστε, το 153 παρακαλώ. Ευχαριστώ που δίνετε το λίγο με Μισελ Αστρουκ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Μεσολαβητών του τομέα της ενέργειας. Θα ήθελα να σας πω ποια είναι η εμπειρία μου που είμαι μεσολαβητής της ZDF Suez. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτά που άκουσα στη συζήτηση. Εκφράζω την ικανοποίηση και τη δική μου και των συναδέλφων μου. Υπάρχουν ατέλειες. Η Μόνικα Κοντιάνς τις ανέφερε. Θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τον καταναλωτή. Και χρειάζεται ε, να δούμε τι γίνεται με τον μεσολαβητή που, δημιουργούν, που θεσπίζουν οι επιχειρήσεις και ποια είναι η σχέση τους που το, με τους μεσολαβητές που τομεακά μπορούν να παίξουν ευρύτερο ρόλο από εμά που είμαστε εντός της Είναι πολύ ποιοτική η δουλειά που γίνεται επί σειρά ετών, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, και έχω δύο κριτήρια με τα οποία τα κρίνω αυτά και αναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα, ο χρόνος. Ο Μπορεί να βρει απάντηση ο καταναλωτής εντός δύο μηνών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το καταφέρνουμε συχνά Δεύτερο κριτήριο σημαντικότατο, επίπεδο ικανοποίηση του καταναλωτού. Διότι θεωρούμε σημαντικό ο διαμεσολαβητή να παίξει το ρόλο του σωστά. Να δημιουργήσει και να βρει λύσει για τα μέρη. Λύσει που να δικαιώνουν τον καταναλωτή στι περισσότερε περιπτώσει. Να σα πω ότι εργαζόμαστε, εξεργαζόμαστε διάφορα είδη διαμεσολάβηση, κυρίω στον ενεργειακό τομέα. Συμμορφωνόμαστε με την οδηγία συνεργαζόμαστε με μεσολαβητή που καθορίζουν τα κράτη-μέλη, συμπροματική προσπάθεια μας για το συμφέρον των καταναλωτών βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Well, Σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια αυτά που βγαίνουν από την πρακτική σας εμπειρία. Ενέργεια και τηλεπικοινωνίες έχουν πράγματι ε, σημαντικά παραδείγματα. Μακάρι να συμβάλλετε και στην δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα ε, τον κύριο που κάθεται στο έδρανο υπαριθμών 196. Παρακαλώ να λάβετε εσείς το λόγο. Και θα ακολουθήσει το 85. Λυπούμε πολύ πολύ για, το, την ανάγκη να σας, ε, να σας ε, αποκαλώ με, τα, με τους αριθμούς αυτούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ο Φεντερίκο Φλαβιάνο από την αρχή για τις τηλεπικοινωνίες ανεξάρτητη υπηρεσία Ιταλική στον τομέα των επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο νόμος μας αναθέτει την αρμοδιότητα να πειθαρχήσουμε και να, τον τομέα και να ελέγχουμε τις διαφορές, να επιλύουμε τις διαφορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ε, λοιπόν, έχουμε απαντήσει στη διαβούλευση τη δημόσια λεπτομερώς και θα ήθελα σε αυτό το βήμα να συνοψίσω τα ισχυρά σημεία της διαδικασίας που ακολουθούμε. 70.000 διαφορές το χρόνο τα τελευταία δύο χρόνια οι περισσότερες διαφορές μέσω της εναλλακτικής μεθόδου επιλύσεως των διαφορών με ποσοστό επιτυχίας και συμφιλίωσης που φτάνουν από 70% μέχρι 95% ανάλογα με τις διαδρομές που επιλέγονται από τον καταναλωτή. Ο πρώτος δρόμος είναι η ε, ισότιμη συνδιαλλαγή. Λοιπόν, και στις, και στις δύο περιπτώσεις και στις επαφές μεταξύ εταιριών και μεταξύ εταιριών και καταναλωτών δίνουμε την ίδια, τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια ποιότητα συνδιαλλαγής και συμφιλίωσης προσ, ε, προσπαθώντας να πετύχουμε και ενθούμε στον δρόμο της υποχρεωτικής συμφιλίωσης. 95% ε, το ποσοστό της επιτυχίας. Οι ενώσεις των καταναλωτών είναι πολύ κοντά στους πολίτες και κινούνται επί τόπου και μπορούν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο. 70% επιτυχία σε περίπτωση όμως την άλλη συμφιλίωση σε, επι, σε, περιφερειακά, σε περιφερειακές επιτροπές των τηλεπικοινωνιών που είναι ανεξάρτητοι φορείς και αυτή. Στην πρώτη και στη δεύτερη υπόθεση που σας ανέφερα, η προσπάθεια συμφιλίωσης και επίσης των διαφορών είναι δωρεάν. Τρίτος δρόμος, ε, στα εμπορικά επιμελητήρια. Ήδη αναφέρθηκαν από την συνάδελφό μας ε, την κυρία Πομπέη. Άλλη ιδιαιτερότητα. Δεύτερη βαθμίδα σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη φάση, δηλαδή διοικητική επίλυση της διαφοράς. Τα συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, ανεξάρτητοι φορεί έχουν περισσότερο περιθώριο να δημιουργούν δίκτυα αυτών των φορέων, των και ανεξάρτητοι φορείς να έχουν αρμοδιότητες και για συναφείς τομείς, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών. Και τέλος, να δημιουργηθεί ένα σήμα ποιότητας που θα μπορεί να τίθεται σε μια συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα είναι ένα σήμα που θα δίνει εμπιστοσύνη, δημιουργεί εμπιστοσύνη στον καταναλωτή και θα ανταποκρίνεται σε ένα υποχρεωτικό δίκτυο σε αυτή την περίπτωση. Όπου εκεί θα εντάσσονται οι φορεί εκείνοι οι οποίοι όταν συμμετέχουν στι συναλλαγέ έχουν το δικαίωμα και βάζουν αυτό το σήμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα έδωσα χρόνο να μιλήσετε γιατί μα είπατε πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και ήταν πλούσιο το υλικό το οποίο μα δώσατε για το τελευταίο αυτό ζήτημα να συστήσω στους συναδέλφους το εξή να σας πω ότι έχει ε, συσταθεί από την Επιτροπή ένας γύρος, ε, ένας, ε, μια ματάργασία υπό την ηγεσία του κ. Άριας για θέματα που αφορούν τέτοια σήματα ποιότητας και ικανοποίησης του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και παρεπιπτόντως Θα δώσω και αργότερα τον λόγο και πάλι στους ομιλητές. Και θα ήθελα να καλωσορίσω την Τζακλίν Μάινερ, που είναι διευθύντρια της ε, πλατφόρμας για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα απαντήσει τα πάρα πολύ δύσκολα ερωτήματα που θα τις θέσω σε λίγο. 85, το αριθμός 85 παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ονομάζομαι ο Χίμπερτ Φαμπρέιμερ και είμαι από την Ένωση Ολλανδικών Επιχειρήσεων, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καταρχάς διοργάνωσε αυτή τη σύνοδο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε και δημοσίευσε το έγγραφο διαβούλευσης στο οποίο φαντάζομαι πολλοί από εμάς εδώ στην αίθουσα μόλις απαντήσαμε. Δεν θα σας δώσω πληροφορίες για το Ολλανδικό σύστημα γιατί ε, ο κύριος Μούρκενς θα μας παρουσιάσει ε, σε λίγο το καλά θεωρώ οργανωμένο Ολλανδικό σύστημα. Να ρωτήσω όμως κάποια, για κάποια πράγματα που περιλαμβάνονταν στο έγγραφο διαβούλευσης. Σε αρκετά σημεία αναφέρονται ποσοστά στο έγγραφο. Τρία μικρά παραδείγματα να σας δώσω. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι 40% των ε, λιανοπολιτών δεν γνωρίζουν καν το ADR. Δεύτερο παράδειγμα, στην παράγραφο υπαριθμών 20 ότι είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά των λιανοπολιτών που χρησιμοποιούν τελικά το ADR. Και τέλος, στην παράγραφο 28 αναφέρεται ότι μόνο το 62% του ADR είναι ανοιχτό σε αλλοδαπούς καταναλωτές. Άρα το λοιπόν, πώς ε, καταλήγουμε σε αυτά τα ποσοστά, πώς τα εξαγάγουμε, γιατί θεωρώ ότι το 62% ή το 40% θα μπορούσε να είναι και καλό αλλά και κακό. Άρα, τι χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε, να εξαγάγουμε αυτά τα στοιχεία. Στις επιχειρήσεις ε, βάζουμε ρεαλιστικού στόχου και ξέρουμε πώς θα του πετυχαίνουμε. Εδώ όμως, σε, αυτό το επίπεδο, πώς μπορούμε να θέσουμε ρεαλιστικού στόχου, Ο πρόεδρο. χαίρομαι που ξεκινάνε οι δύσκολες ερωτήσεις για το πάνελ και τώρα κάποιον που δεν ε, χρειάζεται να τον ε, να του δώσω το λόγο με τον αριθμό του, γιατί τον ξέρω. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέντελτ Μπενισφίλ για, την, ε, για τον έργο της ε, Οικονομικής, Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή σας ε, θα καταρτήσει σχετική έκθεση, γι' αυτό λοιπόν και χαίρομαι που σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Benefit Βίδεσβιλ, δεν μιλώ εξ ονόματος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής εδώ σήμερα. Θα το κάνει αυτό αργότερα ο κύριος Πιγάδο Λής. Να μιλήσω από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Καταναλωτών. Να ευχαριστήσω την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ που ξεκίνησε αυτό το ενδιαφέρον θέμα το οποίο μας αφορά ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει πίστη από πλευράς του καταναλωτή στην ενιαία αγορά και η έλλειψη μιας σωστής ε, μεθόδου αντιμετώπισης των ε, ενστάσεων αποτέλεσε ένα εμπόδιο στο παρελθόν. Το ADR περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία και μου φαίνεται ότι εδώ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το ADR λες και είναι κάτι ενιαίο. Δεν είναι όμως κάτι ενιαίο. Υπάρχουν πολλά είδη ADR γιατί ADR ουσιαστικά είναι οτιδήποτε δεν καταλήγει στο δικαστήριο. Και εδώ να πω ότι υπάρχουν κάποια συστήματα ADR που αξίζουν τον κόπο να τα γνωρίσει ο καταναλωτής. Ίσως τα μοναδικά, ίσως να, σε κάθε χώρο να λειτουργούν διαφορετικά συστήματα. Ως προς τις κατευθυντήριες οδηγίες, να σας πω ότι εγώ έχω εργαστεί στο παρελθόν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και συχνά η διοίκηση μα είπε ότι κοιτάξτε δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριε γραμμές της Επιτροπής επειδή είναι κατευθυντήριε γραμμές μόνο και όχι δεσμευτικέ. Άρα θα ήθελα να έχουμε κάτι πιο δεσμευτικό, να μην έχουμε μόνο κατευθυντήριε γραμμές. Εγώ είμαι από μια χώρα όπου το σύστημα IDR e είναι πάρα πολύ καλά ε, ρυθμισμένο και λειτουργεί πάρα πολύ καλά εδώ και 35 χρόνια. Τα συστήματα αυτά είναι εν μέρη κρατικά και καλύπτουν σχεδόν κάθε τομέα προσφυγών ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν και πολύ καλά συστήματα που έχουν ιδρυθεί από την Δανέζικη Ένωση Καταναλωτών. Για ξενοδοχεία, χρηματοδοτικές υπηρεσίες, οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Και αυτό λειτουργεί πολύ καλά και έχουμε από τη μία πλευρά τους εκπροσώπους ε, των καταναλωτών, τους δικαστές στη μέση και από την άλλη τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα αυτό. Άρα, θα ήθελα να σας ζητήσω να εξετάσετε πρώτα κάποια από τα ήδη υφιστάμενα συστήματα τα οποία λειτουργούν καλά και τα οποία όντω σημαίνουν ότι ο καταναλωτή έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, Μπενεντίτ, και πιστεύω ότι είναι πρακτικό αυτό το θέμα που θίγει. Και φυσικά ανυπομονούμε και για την Δανέσικη Προεδρία μετά την Πολωνική που θα είναι η επόμενη. Υποπτεύομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας αποστείλει και άλλες τέτοιες ιδέες οι οποίες θα αποφέρουν καρπούς ίσως κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας. Ναι, εδώ. μήπω θέλει το λόγο κανένα άλλος συνάδελφος. Σε περίπτωση που δεν θέλει κανείς συνάδελφος το λόγο, θα δώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένου μας. Α, μάλιστα δύο άτομα ακόμα. Ωραία, λοιπόν, δύο σύντομες παρεμβάσει. Και μετά θα περάσουμε και πάλι στο πάνελ. Η κυρία που δεν βλέπω τον αριθμό τη. Γεια σα. Κοντιμάρτυρε από το CCU από την Συνδεμοσπονδία Καταναλωτών και Χρηστών στην Ισπανία. Ήθελα να παρέμβω επειδή αναφέρθηκε ότι υπάρχουν κάποια συστήματα τα οποία λειτουργούν αλλά και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ παλιό σύστημα στην Ισπανία το οποίο εν μέρη μόνο λειτουργεί. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι είναι δεσμευτικό, το οποίο είναι πολύ καλό. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές και αν δεν συμμορφώνεται ο, ο εμπλεκόμενος μπορεί να πάει στο δικαστήριο, αλλά δυστυχώς είναι εθελοντικό. Και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί δεν συμμετέχουν απαραίτητα οι εταιρείε. Εάν ήταν υποχρεωτικό, δεν θα αντιμετωπίζαμε αυτό το πρόβλημα. Και επίση ε, οποιοδήποτε σύστημα θα πρέπει να έχει καλή χρηματοδότηση, το αναφέραμε και στο παρελθόν, αλλά είναι σημαντικό ο υποχρεωτικό χαρακτήρα. Και όπω αναφέρθηκε κάποια από τα συστήματα τα οποία έχουμε και στην Ισπανία, για παράδειγμα στον τομέα του τραπεζικού, στον ασφαλιστικό, δεν λειτουργούν γιατί οι διαμεσολαβητές είναι μέλη του ίδιου του συστήματος εμά. Αυτό δεν είναι διαμεσολάβηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και λυπάμαι που δεν είδα τον αριθμό σας. Έχει ήλιο από πίσω σας, γι' αυτό έχω δικαιολογία. Και άλλη μια κυρία πίσω, τελευταία ομιλήτρια για τον γύρο αυτό. Ευχαριστώ. Μπρίτα Κιόγκεμαν ονομάζομαι, πρόεδρος ε, του Σουηδικού, της Ειδικής Επιτροπής για Επίλυση Καταναλωτών. Θα μιλήσω Σουηδικά, μιας και έχουμε διερμηνία. Thank Σας ευχαριστώ που ήρθατε λοιπόν, που με καλέσατε εδώ πέρα. Στη Σουηδία έχουμε επίσης ένα σύστημα το οποίο υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Το 68 ξεκινήσαμε μάλιστα με το σύστημα αυτό. Έχουμε 21 δικαστές και εγώ είμαι μία εξ αυτών και επιλύονται κάθε έτος πάνω από 10.000 διαφορές. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ε, να ακούμε πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετική η διαμόρφωση του κάθε συστήματος σε κάθε χώρα. Ο κύριος Φρύσο και η κυρία Πομπέη ανέφερα ότι είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να υπάρχει προστασία και της ε, εμπιστοσύνης. Αυτό δεν υπάρχει στη Σουηδία. Δημοσιεύονται τα στοιχεία αυτά. Υπάρχει δημόσια πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και από ό,τι άκουσα πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να μην χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό. Ναι, αλλά στη Σουηδία αποφασίζει ο καταναλωτής κατά πόσον θα καταγγείλει κάποιον. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι στη Σουηδία έχουμε εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, συλλογικέ προσφυγέ. Ω τώρα, το σύστημα αυτό μπορεί να το εφαρμόσει μόνο ο καταναλωτής και ο διαμεσολαβητής. Αλλά την ε, προηγούμενη Δευτέρα ελήφθη μία απόφαση για μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις Υπήρξε ένα ζήτημα για μικρομεσαίες, που έθιξε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ό,τι αφορά τα φορολογικά τους, τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και προτείναμε και πάλι ένα τέτοιο σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας υπενθυμίσατε ότι η λέξη ombudsman είναι όρος σουηδικός που χρησιμοποιείται ευρύτατα και αλλού. Ombudsman διαμεσολαβητή. Καλό. Τη Μόνικα Γκόγιαντς, Φράνσις Ριζόν και την κυρία Πομπέη αν μπορούν να απαντήσουν εν συντομία όσα υπόθηκαν και ο Υπουργός Σέφελτβάη σίγουρα θα θέλει να πει κάποια πράγματα και μετά και οι άλλοι θα θέλουν να πούν κάτι. Έχουμε ένα τέταρτο μέχρι το διάλειμμα για το τσάι. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τέταρτο όμως. Λοιπόν, Μόνικα, εσύ έχεις πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Το τελευταίο σχόλιο σου για το Δημοσιολαβήτη είναι ένας όρος που έχει ιδιαίτερη σημασία στο σκανδιναβικό μοντέλο και που χρησιμοποιήθηκε ποικιλοτρόπως. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο όρος να συνδέεται με συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες. Όσον αφορά τα σχήματα ADR, να τονίσω κάτι που ανηλυμένα υπόθηκε μετά που ακούσαμε τις παρεμβάσεις. Χρειάζεται συμπληρωματικότητα πρέπει να υπάρχει μια μήτρα αποζημίωσης που πρέπει να εφαρμοστεί στους διάφορους τομείς. Αποζημίωση, εξώδικα αποζημίωση, κατόπιν δίκης κλπ. για να έχουν εμπιστοσύνη τελικά στην επίλυση των διαφορών οι καταναλωτές. Περιμένω τα αποτελέσματα α, της αναλύσεως που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση που έγινε. Περιμένω με ανυπομονησία λοιπόν ο κ. φχίζουν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε ακόμα λίγο χρόνο να μιλήσω. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία που αφορούν τη διεξαχθή σας συζήτηση. Καλύτερη γνώση από πλευρά του κοινού, δηλαδή να γνωρίζει το κοινό ότι υπάρχει ένα σύστημα ADR, εναλλακτικό σύστημα επιλύσης των διαφορών. Ο καθένας θα πρέπει να προσπαθήσει και επαγγελματίε, οι δημόσιες αρχές, οι οργανώσει των καταναλωτών θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα προσπάθεια. Η καλύτερη δυνατή διάδοση, διεύρυνση του συστήματο, η δημιουργία εκεί που δεν υπάρχουν συστήματα ADR, όλα αυτά εδράζονται επί ισχυρή πολιτική βουλήσεω των πάντων και σε επίπεδο ενώσεω και σε επίπεδο εθνικό. Απόδειξης αυτού σε κάποιες χώρες, όπω τη Γαλλία, Υπάρχουν υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες στις συμβάσεις, στα συμβόλαια να ενημερώνουν τον καταναλωτή. Και στα ασφαλιστικά συμβόλαια και στους λογαριασμούς των τραπεζών να τους ενημερώνουν ότι υπάρχει μηχανισμός ADR για την επίλυση των διαφορών. Αυτό είναι αρκετά απλό σαν μέσο. Μπορεί να εφαρμοστεί. Όχι επαρκές, αλλά εν πάση περιπτώσει ήδη είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου. Άρα είναι συλλογική η ευθύνη και απευθύνω μια έκκληση εδώ να υπομιστούν όλοι, όλοι τις ευθύνες τους, να μην υπάρχει δισταγμός, ας αναπτυχθεί το σύστημα με κάθε μέσο στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ας ανοίξει ο δρόμος που θα οδηγεί στη γενίκευση χρήσεως του συστήματος, των συστημάτων μάλλον ADR. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πομπέη τώρα έχει το λόγο. Όσον αφορά αυτό που υπόθεση τελευταίες παρεμβάσεις αυτή της επιφύλαξης που υπάρχει ε, είναι κάτι, ε, μάλλον να υπάρχει κάποια εγγύηση για τις επιχειρήσεις σε αυτό το θέμα εμπιστοσύνης. Να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν περισσότερο αυτό το θέμα της και ε, επίλυσης των διαφορών. Έτσι θα μπορούν να φτάνουν πιο εύκολα, αν δεν είναι διστακτικές, στην επίλυση των διαφορών από αυτά που ζήσαμε εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έρχομαι στο άλλο που ήθελα να πω. Γιατί οι εταιρείε δεν χρησιμοποιούν το μέσο αυτό. Διότι δεν το γνωρίζουν, δεν το χρησιμοποιούν. Τουλάχιστον αυτοί, αυτό έχουμε διαπιστώσει. Δεν τον γνωρίζουν. Άρα χρειάζεται επένδυση επί της νοτροπίας όχι μόνο στον υποχρεωτικό χαρακτήρα που προανέφερα στην προηγούμενη παρέμβαση, αλλά μέσω επικοινωνίας, ενημέρωσης. Εμείς σαν επιμελητήρια προσπαθούμε, επενδύσαμε επ' αυτού τα τελευταία χρόνια, να επικοινωνήσουμε, να καταλάβουν οι επιχειρήσεις μας περί τι πρόκειται, τι είναι η διαμεσολάβηση, ποια είναι τα ωφέλη, τι μπορούν να βρουν στα εμπορικά επιμελητήρια, ποιος είναι ο διαμεσολαβητής, τι είναι η διαμεσολάβηση. Αυτό είναι σημαντικό πέρασμα, αν θέλετε, ένα βήμα που πρέπει να γίνει. Τελευταίο θέμα, η ενώση των καταναλωτών. Ο συνάδελφο τη Αρχή για τι Τηλεπικοινωνίε αναφέρθηκε στο θέμα. Είναι σημαντικό αυτό. Στην ιστορία το δοκιμάσαμε. Είναι εμπειρία σημαντική και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Στη χώρα μα ήταν πρώτη σε αυτό το τομέα που εφάρμοσαν τη μεσολάβηση και την συνδιαλλαγή και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτό και να εξακολουθούν να αξιοποιούνται αυτές οι προσεγγίσεις και αυτές οι λύσεις. Αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευρύν, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Ε, αφού και η παρουσιάστηκε, ας πούμε, η της, ε, της ε, διασκέψεως. Πάντως, όπως είπαν ορισμένοι ομιλητές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία μηχανισμών σήμερα στις διάφορες χώρες μέλη και διαφορετική ποιότητα απόδοσης των διαφόρων συστημάτων. Υπάρχουν πληροφορίες για τα συστήματα αυτά Υπάρχουν και πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει τα θεσμικά όργανα για να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα των διαφόρων μηχανισμών που υπάρχουν σε διάφορες χώρες μέλη. Σωστό είναι να διατηρηθεί μια ευκαμψία, όπως λέχθηκε πριν. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα τα οποία επανέρχονται και φαίνεται να είναι σχετικά εύκολο να αναλάβει κανείς δράση, όπως η έλλειψη ενημέρωσης, έλλειψη γνώσης, το θέμα της εμπιστευτικότητας, στην ε, Σουηδία αυτό το λεγόμενο naming and shaming φαίνεται πως λειτουργεί καλά ώστε να αναγκάζει τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων της εναλλακτική διευθέτησης διαφορών. Αυτό που προκύπτει από τις διάφορες παρεμβάσεις είναι πάντως, αυτό προκύπτει, είναι η ανάγκη ανάληψης δράσης και αυτό θα πρέπει να είναι και το θέμα και για την επόμενη ε, διάσκεψη. η γειτόνισσα μου δίπλα θα προεδρεύσει της επόμενης, ε, το επόμενο τμήματος της διάσκεψης. Εσείς κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δώσατε να ακούσω ε, τις διάφορες παρεμβάσεις για την ποικιλία των μηχανισμών εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ευνοϊκών προϋποθέσεων που ήταν και το πρώτο που είπα στην παρέμβασή μου αλλά άκουσα και πολλές ερωτήσεις και παρατηρήσεις και με ενισχύει στην άποψή μου αυτό ότι δηλαδή χρειάζεται ένα, ένα, ένα, ένα πλαίσιο ευνοϊκών προϋποθέσεων που να διευκολύνει την χρήση των συστημάτων ADR. Θα κάνω δύο σχόλια για θέματα που νομίζω έχουν σημαντική, ε, ε, σημαντικό ρόλο εδώ. Αφενό είναι η αύξηση της ενημέρωσης, της γνώσης για την ύπαρξη των συστημάτων εναλλακτική διευθέτηση διαφορών. Άκουσα πολλού να παραπονούνται για την έλλειψη τη ενημέρωση αυτή. Πρέπει να κάνουμε κάποια περισσότερη, κάποια μεγαλύτερη προσπάθεια από το να λέμε απλώ στον κόσμο ότι υπάρχει το σύστημα αυτό. Πρέπει, χρειάζεται μια πιο συστηματική προσέγγιση. Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει. Το άλλο που έχει μεγάλη σημασία είναι να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των μηχανισμών εναλλακτικής διευθέτησης διαφόρων. Άκουσα τις διάφορες ποικίλε εκφάνσεις. Είναι σημαντικά βέβαια αυτά για τους καταναλωτές, αλλά και για τους εμπόρους, για τις επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο το ADR να διαθέτει μια ποιότητα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Να υπάρχει δηλαδή value for money όπως λένε στα αγγλικά. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τα συστήματα εναλλακτική διευθέτησης διαφορών θα κοστίσουν κάποια χρήματα. Θα χρειαστεί λοιπόν να γίνει κάποια επένδυση σε τα συστήματα αυτά αν θέλουμε να έχουμε καλές υπηρεσίες. Ε, Επειδή εδώ επιθυμώ να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα. Εγώ είμαι στο Υπουργείο Οικονομίας. Βλέπω λοιπόν και τις δύο πλευρές, όχι μόνο των καταναλωτών, αλλά και αυτών που προσφέρουν υπηρεσίες. Που παράγουν δηλαδή το προϊόν αυτό. Χρειάζεται εξέταση και των δύο πλευρών. Ε, οι καλοί μηχανισμοί εναλλακτική διευθέτηση διαφορών πρέπει να αποβαίνουν προ όφελο και των δύο πλευρών. Πολλοί βέβαια ρίχνουν ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των καταναλωτών και, και σωστά κάνουν. Αλλά αυτό ήθελα να πω, ε, να σας παρακαλέσω όλες και όλους να εξετάσετε και τις δύο πλευρές, γιατί όπως είπα πρέπει να είναι αμοιβαία υποφελές το σύστημα και για τις δύο πλευρές της εξισώσεως. Κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το πρώτο μέρος της Σας Ευχαριστώ όλες και όλους όσοι παρενέβητε. Θα διακόψουμε για να πιούμε ένα καφέ. Ο Τζον Ντάλι, η Γενική Διευθύντρια μάλλον του Τζον Ντάλι, επειδή είναι αρμόδια και για την υγεία, έχει προσφέρει φρούτα. Όχι μόνο καφέ λοιπόν, αλλά και άλλα εδέσματα που θα σας δώσουν δύναμη και για την επόμενη και το επόμενο μέρος. Θα ήθελα να ε, χειροκροτήσουμε τους τελευταίους ομιλητές μας. Uh, thank you everybody for being back so punctually. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην ώρα σας. Χαίρομαι που απολαύσατε τα φρουτάκια. Και όταν φεύγετε παίρνετε ένα πορτοκαλάκι, ένα μιλαράκι για να θυμόσαστε αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση. Θα δώσω το λόγο για το επόμενο τμήμα της συζητήσεως στη Jacqueline Μάινερ που θα διευθύνει την συζήτηση που ακολουθήσει, διευθυντρία για θέματα υποθέσεων καταναλωτών ε, στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΚΟ. Της δίνω το σφυράκι και ξεκινάμε αμελητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή τη ε, διάσκεψη και όλους σας. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς με την ανταπόκριση που βλέπουμε και σήμερα το απόγευμα, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Είχαμε λάβει 200 απαντήσεις τελευταία φορά που μετρήσαμε, αυτό και, ε, και ε, διπλασιάζονται <laughs> μάλλον ε, κάθε μέρα και μπορεί να φτάσουμε 400 αύριο. Θα έρθουν πολλές ακόμα. Σκοπός τώρα του τμήματος αυτού της συζητήσεως είναι να δούμε ποιο είναι το μέλλον όσον αφορά το ADR e ή την εναλλακτική διαθέτηση των διαφορών, φίλης των διαφορών. Στο πρώτο τμήμα δημιουργήθηκε η βάση για την συζήτηση που ακολουθήσει τώρα. Το είπε και Εύελιν. Αυτό που διαφάνει από την πλουσιότατη και άκρως ενημερωτική συζήτηση ήταν η μεγάλη επικοινομορφία που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις λύσεις ADR, προσφορά, πώς λειτουργούν, πώς γίνονται αντιληπτέ από επιχειρήσεις και καταναλωτές. Βασική μας πρόκληση, πιστεύω, στο μέλλον είναι να εξασφαλίσουμε ότι διατηρούμε τα καλά στοιχεία και αυτά που πηγαίνουν καλά τώρα. Αν κάτι δεν έχει βλάβει, μη το μαστορεύεις όπως λέμε. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν ό,τι λειτουργεί να τα αφήσουμε. Να το διατηρήσουμε. Κάποιοι είπαν ότι όμως υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις αρχές, βασικά κριτήρια που θα πρέπει να τα ακολουθεί κάποιο σύστημα EDR που είναι άξιο, αντάξιο του ονόματός τους. Πρέπει να συζητήσουμε ποια θα είναι τα κριτήρια και υπάρχουν ένα-δύο δύσκολα ερωτήματα. Τα είδαμε, εφήγησαν στην προηγηθή σας συζήτηση, δηλαδή το να ανήκει κανείς σε κάποιο τέτοιο μηχανισμό θα πρέπει να ανήκει α, ε, ε, εθελοντικά, υποχρεωτικά οι αποφάσεις του συστήματος ADR θα είναι δεσμευτικές όσον αφορά τα μέρη που έχουν προσφύγει σε αυτό ή όχι. Η ευαισθητοποίηση πώς αυξάνεται όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των εμπορευομένων. Ποια είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα που ίσως προκύψουν σε διασυνοριακό επίπεδο. Η γλώσσα είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που θα ανακύψουν σε διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Και κάτι άλλο που δεν έφυγε στη συζήτηση. Οι ιδιαιτερότητε του online, τη της διαφορών online υπάρχουν. Πρέπει να επιλύσουμε ιδιαιτερότητε εκεί να βρούμε ποιε είναι. Αυτές είναι οι ερωτήσεις και ελπίζω να βρουν κάποιες απαντήσεις ε, στα επόμενα 90 λεπτά. Έχω πολλούς διακεκριμένους ομιλητές που θα ξεκινήσουν ε, τη συζήτηση με παρεμβάσεις. Θα δώσω το λόγο στην Σάντρα Κανιέτε, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής ΙΜΚΟ, που είναι η συγγήτρια για την πολύ σημαντική γνωμοδότηση για τη διακυβέρνηση στην ενία αγορά, όπου εκεί ε, αναφέρθηκε εκτενώς το θέμα αυτών των αλλακτικών μηχανισμών περιουσίων διαφορών. Η EDR, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, η κυρία Κανιέτε, ευχαριστώ. Διακεκριμένοι συνάδελφοι, συμμετέχοντες σε αυτή την συζήτηση. Σήμερα ενέκρινε τις εκθέσεις η Επιτροπή μας όσον αφορά την ενιαία αγορά και την πράξη για την ενιαία αγορά και είχα την τιμή να επισεργαστώ την έκθεση για την διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά. Πολύ καλές ήταν συζητήσεις που έλαβαν χώρα βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια ε, δράση που είχε προτεραιότητα ενεκρίθη από, όλα τα, από όλες τις πολιτικές ομάδες. Αναφέρομαι στου μηχανισμού, εναλλακτικού μηχανισμούς επιλύσεων διαφορών, ADR, που είναι μέσα στι πέντε προτεραιότητε για δράση όσον αφορά τη διακυβέρνηση τη νέα αγορά. Προσβλέπουμε στι προτάσει νομοθετικού περιεχομένου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ADR. προτάσει που επιβληθούν φέτος. Πρέπει γρήγορα να εγκριθούν σχετικέ προτάσει. Υπάρχουν πτυχέ των ευρωπαϊκών ADR, του ευρωπαϊκού ADR μάλλον, που θα ήθελα να τονίσω κατά τράποψή μας, ταχεία και αποτελεσματική προσφυγή σε μηχανισμούς διευθετήσεως των διαφορών εξώδικα είναι κάτι εποφελές και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Γιατί για τις επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις όλος ιδιαίτερος συχνά βρίσκονται σε παρόμοιες θέσεις με μεγάλες, μεγάλους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Όπως και οι κατανοτέ άλλωστε. Χρειάζεται καλύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Πιστεύει η Επιτροπή ότι ένα EDR ευρωπαϊκό πλήρες και σχετικό πλαίσιο που θα καλύπτει διαφορές εθνικές και διασυνοριακές είναι κάτι που απαιτείται. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το τμήμα που αυξάνεται σε μέγεθος των αγορών online και η διαθεσιμότητα των ADR θα πρέπει να γνωστοποιείται καλύτερα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποχρεωθούν να καταβάλουν προσπάθειες προς ενημέρωση των καταναλωτών όταν συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα ADR και όταν δεν συμμετέχουν. Αποτελεσματικός τρόπος για να ενημερώνουν για τη θεσιμότητα ADR είναι μέσω εργαλείων online, όπως βάσει δεδομένων ευρωπαϊκή online όπου κάθε καταναλωτής μπορεί να δει συμμετέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση σε σύστημα EDR ή όχι. Ποιος είναι ο ακριβής μηχανισμός. Ποιοι είναι οι κανόνες. Άρα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το EDR. Και θέλουμε γρήγορα να υιοθετηθούν μέτρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ ε, σε αυτά που μας είπατε και σύντομοι και πλήρης. Ο κ. Λόικ Αρμό, Γενικός Διευθυντής για βιώσιμη ανάπτυξη, σχέση με τους καταναλωτές και δημόσια θέματα, του φορέα του που εδρεύει στο Παρίσι, συμμετείχε ενεργά στο έργο του Μέντεφ, που είναι η Γαλλική ο Γαλλικός Φορέας για τη Βιομηχανία, για τη διαμεσολάβηση ή mediation γαλλιστή, ADR, θα μας πει τι γίνεται στη Γαλλία. Και πώς οι γαλλικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στη δημιουργία του ADR στη Γαλλία. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Το θέμα αυτό το λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά στην ΜΕΝΤΕΦ στη Γαλλική Ένωση Επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος να πείσουμε τους καταναλωτέ και τους προμηθευτές να χρησιμοποιούν την διαμεσολάβηση όταν δεν βρίσκουν λύσεις ε, για τις διαφορές είναι να δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα και τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Δεν θα, δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσαμε. Λίγα λόγια όμως να πω ότι καταρχάς ε, μετράει πάρα πολύ ταχύτητα. Δύο μήνες, για παράδειγμα, αντί για χρόνια δικαστικών διαδικασιών. Κανένα κόστος για τον καταναλωτή, χαμηλό κόστος. Το απόρριτο της ε, διαδικασίας. Επειδή υπάρχει και ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος, υπάρχει σωστή πρόσβαση και για τα δύο μέρη στη σωστή τεχνική και νομική ε, αρρωγή. Τα θετικά αποτελέσματα στη Γαλλία φτάνουν μέχρι και 90% των περιπτώσεων. Επίσης, η διαμεσολάβηση μπορεί να παρέχει μια δίκαιη λύση που θα ωφελήσει και τους καταναλωτές, ενώ η εφαρμογή των νομικών διατάξεων μπορεί να μην αποβεί προς όφελος του καταναλωτή. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό για τους παρόχους, ότι η διαμεσολάβηση προστατεύει και την επιχειρηματική αυτή σχέση. Και τέλος, να τονίσω την σημασία της ελεύθερης επιλογής. Και οι δύο πλευρές μπορούν ανα πάσα στιγμή να αποσυρθούν και να αποτανθούν στα δικαστήρια σε περίπτωση που το θεωρήσουν προτιμητέο. Η διαμεσολάβηση δεν αντικαθιστά την ε, δικαστική διαδικασία. Απλά αποσκοπεί στο να την καταστήσει Και αυτό έχει διαφορά. Γιατί δουλεύουμε τόσο πολύ για το ADR στην ΜΕΝΤΕΦ στη Γαλλία, γιατί θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικά παρόμοια συμφέροντα. Η ΜΕΝΤΕΦ ε, θέλει να κερδίσει την ε, εμπιστοσύνη των ε, επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην διαμεσολάβηση. Τι κάνουμε λοιπόν και ποιος θεωρούμε ότι είναι ο μελλοντικό τρόπος διαμόρφωσης του ADR. Εμάς μας απασχολούν τρεις πρωτοβουλίες. Καταρχάς, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση των επαγγελματιών και των ε, καταναλωτών. Κατά δεύτερον, θέλουμε να δίνουμε εγγυήσει στον καταναλωτή για την ποιότητα της διαμεσολάβησης. Κατά τρίτον, θέλουμε να διευρύνουμε τη γεωγραφική προσφορά και την τομεακή προσφορά του IDR. Κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα θεωρούμε ότι όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι, διαδραματίζουν το ρόλο τους. Οι επαγγελματίες, για τις επαγγελματίες τον Μάιο του 2009, η ΜΕΤΕΦ δημοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό για την διαμεσολάβηση για να συμβάλλει στη διεύρυνση των εξειδικαστικών αυτών λύσεων. Επίσης, δημιουργήσαμε ένα φόρουμ των διαμεσολαβητών που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις διαμεσολαβήσεις για να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2010 η ΜΕΔΕΦ ξεκίνησε έναν ε, κόμβο στο διαδίκτυο για να παρέχει μεταξύ άλλων ε, πληροφορίες για τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Ωστόσο, θεωρούμε ότι και οι αρχές, οι κρατικές έχουν το ρόλο τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε κρατικό επίπεδο. Στη Γαλλία, το Εθνικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2007 με ομόφωνη απόφαση των ενώσεων καταναλωτών ενέκρινε μια γνωμοδότηση για την διαμεσολάβηση και για το ADR και τον Οκτώβριο του 2010 συστάθηκε μια επιτροπή διαμεσολάβησης η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2011. Θεωρούμε ότι και οι κρατικοί φορείς έχουν σημαντικό ρόλο ως προς την ενημέρωση του καταναλωτή. Τέλος, θα είναι σημαντικό να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα, να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Πιο πολλές ε, εγγυήσεις τώρα και τον καταναλωτή. Έχουμε δημοσιεύσει τις αρχές ε, της αμερόληπτης διαμεσολάβησης βάσει της απόφασης ε, που έλαβε το Εθνικό Συμβούλιο Κατανάλωσης το 2007 σε ό,τι αφορά τα θέματα αμεροληψίας. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να συγχαίουμε την ανεξαρτησία με την αμεροληψία, γιατί η αμεροληψία σημαίνει εξαρτησία στο μυαλό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να αναφέρει κάθε φορά στον πρόεδρο της Επιτροπής. Πρέπει να έχει χρηματοδότηση, δεν μπορεί να λαμβάνει αποζημίωση για την διαμεσολάβηση, την κάθε διαμεσολάβηση και θα πρέπει φυσικά να μην εμπλέκεται σε σύγκρουση συμφερόντων. Αυτές οι αρχές δημοσιεύτηκαν το 2010 από τη ΜΕΝΤΕΦ. Για να διευρυνθεί τώρα το πεδίο προσφοράς, θα ήθελα να πω ότι έχουμε διάφορους ε, κλάδους και βιομηχανίες ε, στην Γαλλία που καλύπτονται ήδη από διαδικασίες διαμεσολάβησης, μα τράπεζες, ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τεχνολογικές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες και άλλες. Και πρόσφατα διευρύθηκε και στις οικοδομές και στην παροχή υδάτος, στις ενεργειακές εταιρείες Έχουμε και στην EDF και στην CDF Suez και σε franchise, εταιρείε franchise. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το σύστημα με γεωγραφικά δίκτυα προκειμένου να καλύπτονται καταστάσεις όπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα είχαν ενδεχομένω κανένα συγκεκριμένο σύστημα διαμεσολάβησης στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. <clears throat> Το τελευταίο που είπατε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τρόποι με τους οποίους προσπάθησε να θέσει υπόψη και των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών η ΜΕΝΤΕΦ την ύπαρξη των μηχανισμών διαμεσολάβησης ένα σύστημα που έχει εδαφική βάση και που καλύπτει τις μικρές κυρίως εκείνες επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στο κεντρικό σύστημα εναλλακτική διευθέτηση ε, διαφορών. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των τομέων εκείνων που είναι κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, όπου δραστηριοποιούνται μεγάλες επιχειρήσεις με πολύ αυστηρή νομοθετική ρύθμιση και προχωρούμε μετά στον τομέα του λιανικού εμπορίου, όπου συμμετέχουν πολλέ μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, με πολύ λιγότερη νομοθετική ρύθμιση στην πραγματικότητα, και όπου το ADR στον πρώτο τομέα έχει μεγάλη διάδοση, στον δεύτερο τομέα πολύ λιγότερο. Είναι ένα θέμα αυτό νομίζω το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Θα ακολουθήσει τώρα πάλι ένας ευρωβουλευτής ο κύριος Ραφαέλε Μπαλντασάρε είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα ωφέλη της εξοδικαστικής επιλύσεως των διαφορών είναι πάρα πολλά και συμφωνούμε. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Μειώνεται επίσης και μειώνονται και οι υποθέσεις που δικδικάζονται που σε κάποιες χώρες παθολογικά, είναι παθολογικά υψηλός ο αριθμός τους και επιτρέπεται και μια γρήγορη ε, λύση και με χαμηλό κόστος. Λοιπόν, είναι πολύ περιορισμένη η γνώση αφορά αυτά τα συστήματα και αυτό συνεπάγεται την ανάγκη οι καταναλωτές ε, να, να ξέρουν το θέμα αυτό που τους βοηθάει να αποφύγουν το κόστος που έχει να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Άρα πρέπει να γνωστοποιηθεί αυτό το σύστημα επιλύσεως των ε, διαφορών μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων. Γι' αυτό οι ενώσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων μπορούν να συμβάλλουν και με πολύ σημαντικό τρόπο. Όσον αφορά τους καταναλωτές, επί παραδείγματι, European Consumer Centers Network, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τα network, τα δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν τράπεζες δεδομένων για να εντοπίζονται οι δύο προσφυγής και κατά κάποιο τρόπο να βυθίζουν τις υποθέσεις και να αφαιρούν τους φραγμούς, κυρίως τους γλωσσικούς, για την υλοποίηση των δικασιών. και, θα, και συνδέεται η αποτελεσματικότητα των ADR από το σωστό νομικό σύστημα και έτσι η, αν ήταν το δικαστικό σύστημα λογικό και το νομικό θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για να ε, λύνει τις διαφορές σε πιο εύλογο χρονικό διάστημα. Και να, μην, ε, να μειωθούν εκείνοι που καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για να εκμετάλλευονται την καθυστέρηση επιλύσης των διαφορών για να κολλησιεργούν. Εάν έχει κανεί διαμεσολαβητή καλά προετοιμασμένο και κατάλληλου μηχανισμού, μπορεί να λυθεί σωστά το θέμα. Χρειάζονται αυστηροί κανόνε για την επιλογή εκείνου που θα είναι υπεύθυνοι για τη λύση και επαρκέ μορφέ δημοσίου ελέγχου όσον αφορά την ποιότητα των πανεχομένων υπηρεσιών. Πέρα από τι βελτιώσει του δικαστικού συστήματο και του νομικού συστήματο, θα πρέπει να διαδοθεί το σύστημα να χρησιμοποιούν τα μέρη περισσότερο τις διαδικασίες της επιλύσεως των διαφορών, εναλλακτικών μεθόδων ε, επιλύσεως των διαφορών EDR. Γι' αυτό Θα πρέπει να αξιολογεί ο δικαστής αν δεν έχει επιληθεί διαφορά από το ADR e και τελικά προσφύγουν στη δικαιοσύνη ο δικαστής να το λαμβάνει αυτό υπόψη του. χρειάζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για τα EDR και μπορεί να είναι συμπληρωματική λύση και εναλλακτική λύση στις δράσεις συλλογική ε, προσφύγης. Κυρίως στις χώρες εκείνες που μόλις πρόσφατα και στην Ευρώπη ξεκίνησαν την πολιτική συζήτηση για τη σκοπιμότητα εγκρίσεως τέτοιων δράσεων, των περίφημων class actions. Άρα θα πρέπει να δούμε και όλα κλασικά μοντέλα γιατί όσον αφορά την παρέμβαση τρίτου στη διαμεσολάβηση. Διερευνώντας φιλικές λύσεις που μπορούν να διαπραγματευτούν μεταξύ τους τα μέρη. Το, το μοντέλο το ισο, ισότιμης επιλύσεως των διαφορών ίσως να είναι εναλλακτική μέθοδος για τη συμφιλίωση χωρίς την παρέμβαση τρίτων μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων μερών. Εάν υπάρχει συμφωνία βάσει πρωτοκόλου μεταξύ ενώσεως καταναλωτών και επιχειρήσεων όπου τα μέρη δεσμεύονται να θέσουν επιτροπή την επίλυση διαφορών, αυτό επιτρέπει να ε, επιτευχθούν διάφορα ωφέλη. Σε αυτό το μοντέλο οι επιχειρήσεις μπορούν αποτελεσματικά να επιλύουν επωφελώς πολλές διαφορές που παράγονται διαδοχικά. Ταυτόχρονα το σύστημα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας και εκπροσώπησης των καταναλωτών ο καταναλωτής που εκπροσωπείται στην Επιτροπή της Ενώσεως δεν υπόκειται σε αυτή την ε, ασυμμετρία όσον αφορά την ενημέρωση και τη δυσχερή θέση που έχει έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. δυσμενή θέση. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, last but not least, τα συστήματα επιλύσεως των διαφορών, τα εναλλακτικά συστήματα επιλύσεως των διαφορών θα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση ε, της αναπτύξεως του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δείκτες αναπτύξεως του εμπορίου του ηλεκτρονικού είναι πολύ χαμηλοί. 7% μόλις του διασυνοριακού εμπορίου γίνεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαρτάται από την εμπιστοσύνη που έχει ο καταναλωτής στο σύστημα και πόσο αποτελεσματικό είναι το δίκαιο που εφαρμοστεί εκεί. Χρειάζονται δικασίες γρήγορες, φτηνές για τη διαχείριση των παθολογικών σχέσεων μεταξύ καταναλωτού και πολιτού και εταιρεία. Είναι θεμελιώδες στοιχείο αυτό για την καλή, καλό αποτέλεσμα των σχέσεων και την σύναψη των συμβάσεων. Και τα μέτρα σε δίκτυο είναι σημαντικές μέσω υπολογιστού να μπορεί χωρίς να μετακινείται ο καταναλωτής να απευθύνεται προς την εταιρεία ή στην ένωσή του και να ξεκινά μια διαδικασία ADR. Χρειάζεται λοιπόν συμπληρωματικότητα των συστημάτων των ADR να συνοδεύουν και να συμπληρώνουν άλλα συστήματα που αναλύονται στο Κοινοβούλιο. Έτσι θα προστατεύεται ο καταναλωτή. Η προστασία θα είναι υψηλού επίπεδου και θα υπάρχει και νομική κάλυψη σε δυσονικό επίπεδο. Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινό εργαλείο, έστω και με δυνητική ευχέρεια, ε, που θα διέπει το δίκαιο ε, των συμβάσεων που συνάπτονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Um, Σας ευχαριστώ. <clears throat> Είπατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Θα έλθω σε λίγα από αυτά. Πρώτα, η σχέση μεταξύ της εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών και των δικαστικών διαδικασιών. Βεβαίως υπάρχει και η διασύνδεση που ανέφεραν και προηγούμενα άλλοι ομιλητές ανάμεσα στο ADR και στις συλλογικές ε, ε, αγωγές για αποζημίωση. Τι γίνεται όμως με, τις, ε, με τον χρόνο παραγραφής. Αναστέλλεται η πάροδος του χρόνου παραγραφής όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Μπορώ τώρα να προχωρήσω στον επόμενο ομιλητή μας που είναι ο Πέτερ Φοχ Κνούτσεν, ε, είναι διευθυντής του Δανικού Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει και εμπειρία και διαμεθοριακής διαμεσολάβησης δηλαδή ε, χορηγεί συμβουλές σε καταναλωτές και όταν έχουν θέματα διαμεθοριακά και ελπίζω ότι θα μας ε, δώσει κάποια από τα, θα μας ε, θέσει υπόψη κάποια από τα μαθήματα της εμπειρίας του. Έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διαμεθοριακές διαφορές όταν μιλούμε για την ανάπτυξη μηχανισμών εναλλακτική διευθέτηση διαφορών. Το δίκτυό μας έχει σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Το 2010 λάβαμε περίπου 32.000 καταγγελίες από ε, καταναλωτές και 60% είχαν σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πολλές από τις καταγγελίες αυτές αντιμετωπίστηκαν ήδη από το ECC, αλλά σε 13.000 υποθέσεις ο καταναλωτής και η χώρα του καταναλωτού ζήτησαν αρρωγή από την χώρα Τη επιχείρησης και πάλι στι μισέ από αυτές τις υποθέσεις είχαμε ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα περισσότερα, οι περισσότερες καταγγελίες που λάβαμε αναφέρονταν σε βασικά προβλήματα, 30% περίπου σχετικά με το προϊόν, είτε <clears throat> με ελαττωματικά προϊόντα, είτε με τον τρόπο που ε, έγινε η παραγγελία. Επίσης, η παράδοση του προϊόντος ήταν ένα 20%. Απλό πρόβλημα που ωστόσο προκαλεί πολλά προβλήματα σε πολλούς καταναλωτές. Ή αγοράζετε ένα εισιτήριο για μια συναυλία σε άλλη χώρα, πληρώνετε το εισιτήριο, μετά αγοράζετε το εισιτήριο του αεροπλάνου, κλείνετε δωμάτιο στο ξενοδοχείο και εν τέλει δεν σας έρχεται ποτέ το εισιτήριο της συναυλίας. Έτσι λοιπόν όχι μόνο δεν έχετε το εισιτήριο της συναυλίας το οποίο επιθυμούσατε, αλλά έχετε και έξτρα δαπάνες, κάνει που ήταν περιτές εν τέλει. Το ECC μπόρεσε να λύσει πολλές από τις υποθέσεις αυτές, για τις μισές περίπου. Είναι καλό αυτό, διότι δεν έχουμε βεβαίως ε, καμία εξουσία καταναγκασμού, αλλά υπάρχει και το άλλο μισό υποθέσεων που δεν μπορέσαμε να λύσουμε, κυρίως λόγω της έλλειψης συμμετοχής των εμπόρων για αυτό το δεύτερο μισό των καταγγελιών οι καταναλωτές αφήνονται στην μοίρα τους όταν μιλούμε για διαμεθοριακές υποθέσεις. Η Κομισιόν μιλεί για κλείσιμο κενών για θέματα ADR θεωρώντας ότι τα κενά αυτά είναι η μικρή εκείνη τομή που δεν υπάρχει ακόμα το ADR αλλά σε ό,τι αφορά το διαμεθοριακό ADR είναι περίπου το 90% 95% που σημαίνει ότι μόλις 5% εμείς στο δίκτυο ECC μπορούμε να ε, υποβάλουμε τις υποθέσεις αυτές σε ένα υφιστάμενο μηχανισμό εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών, διότι απλώς δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί. Οι καταγγελίες προέρχονται κυρίως από υποθέσεις Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου οι συνάδελφοί μου μπόρεσαν μόνο 40 υποθέσεις να θέσουν υπόψη του ADR το 2007 και 8. Δεν μιλώ για 40%, μιλώ για 40 υποθέσεις σε δύο χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ένα μέγα κενό. Οι καταναλωτές που έχουν δυσάρεστη εμπειρία γιατί κανείς δεν τους βοήθησε θα πούν και στον περιβάλλον τους και στο οικείο, στο οικείο και φιλικό περιβάλλον τους την εμπειρία τους αυτή και αυτό εξηγεί την επιφυλακτικότητα του κοινού. Για να γίνει τώρα η εσωτερική ενιαία αγορά πραγματικότητα για τους καταναλωτές πρέπει να αναπτυχθεί ο διαμεθοριακός μηχανισμός εναλλακτική διευθέτησης διαφορών. Και αυτό θα πρέπει να μπορεί να γίνει και επιγραμμικά. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η γλώσσα. Η γλώσσα την οποία μπορεί να υποβληθεί ε, η καταγγελία. Υπάρχουν βέβαια διάφορα μοντέλα που μπορεί να επιλέξει κανείς. Γνωρίζω ότι γίνεται σχετική έρευνα για να υπάρξει ένα κοινό ADR για έναν τύπο καταγγελιών και μάλιστα να υπάρξει όχι μόνο ευρωπαϊκός ADR αλλά και παγκόσμιος. Υπάρχει και πρωτοβουλία ε, και κυβερνήσεων αλλά και ιδιωτικών οργανώσεων για να υπάρξουν αυτές οι ρυθμίσεις. Αν όμως είχαμε μηχανισμό εναλλακτική διευθέτηση διαφορών για διαμεθοριακές διαφορές, το προφανές, απο... το πλεονέκτημα θα ήταν ότι θα πρόσφερε ε, επιπλέον ε, δυνατότητες στους καταναλωτές για να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει. Είμαστε αναγκασμένοι λοιπόν να πούμε σε 50 έω 60% των καταναλωτών που ακόμα δεν έχουν κάνει αγορές επιγραμμικά, τι μπορούν να κάνουν σε περίπτωση προβλημάτων. Μπορούμε να τους πούμε λοιπόν ότι έχουν κάποιον να απευθυνθούν εφόσον αντιμετωπίσουν προβλήματα στις ε, συναλλαγές τους αυτές. Και να μην περιοριστούν μονάχα στην καλή βούληση του παρόχου. Θα έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές ε, να λάβουν αυτά στα οποία έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά τη γνώμη μου αυτό θα προσφέρει πολύ περισσότερα στην ε, ανύψωση του επίπεδου προστασίας των καταναλωτών και στις διαμεθοριακές ε, υποθέσεις. Διότι χωρίς την δυνατότητα επιβολής των κανόνων, οι ίδιοι κανόνες δεν έχουν μεγάλη αξία. Το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι θα πρέπει η συμμετοχή για τις επιχειρήσεις να είναι υποχρεωτική ή τουλάχιστον να καταστεί δυνατόν στον μηχανισμό εναλλακτική διευθέτηση των διαφορών να μπορεί να αναλάβει δράση ανεξαρτήτως του αν επιθυμεί ή όχι να συμμετάσχει ο επιχειρηματίας. Μέχρι τώρα στα έξι χρόνια που έχω εργαστεί στα θέματα αυτά ποτέ δεν άκουσα κάποιον επιχειρηματία που να θέλει εθελοντικά να συμμετάσχει. Άρα εθελοντικός ADR σημαίνει για μένα έλλειψη ADR. Η συμμετοχή λοιπόν των εμπόρων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για θέματα διαμεθοριακών διαφορών. Εάν δηλαδή θέλουμε πραγματικά να προκαλέσουμε κάποια διαφορά υπέρ των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βεβαία ότι θα θυμηθούμε πολλά από τα όσα είπατε ε, στην παρέμβασή σας που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Θα προχωρήσουμε αμέσως γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι ομιλητές έχουν πολλά να πούν θα προχωρήσουμε στον τελευταίο ευρωβουλευτή που είναι ο κύριος Κρόιτσμαν της Επιτροπής Προστασίας Καταναλωτών και σκιώδης εισηγητής για την έκθεση Γκερέρο Κάμπος για την ενιαία αγορά υπέρ των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή εκδήλωση δείχνει ότι μπορούμε να λάβουμε σημαντικά μαθήματα από όλες τις παρεμβάσεις Έχουμε ζητήσει να τεξαχθεί μελέτη για διαμεθοριακά συστήματα ADR, η οποία δυστυχώς δεν πρόλαβε να συνταχθεί εγκαίρως για τη σημερινή διάσκεψη. <clears throat> Θα την έχουμε σε δύο μήνες περίπου και την αναμένω με ενδιαφέρον. Και οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα θέματα των συστημάτων ADR να μπορέσουν να διαμορφωθούν και ιδίως να ωφεληθεί ο καταναλωτής θα θέσω υπόψη σας ορισμένες προτάσεις, διότι το θέμα είναι πώς μπορούμε να εξελίξουμε περαιτέρω τους μηχανισμούς αυτούς. Σε όλες τις παρεμβάσεις έθεσαν οι παρεμβαίνοντες το θέμα της γνώσης ή της έλλειψης γνώσης σχετικά με την ύπαρξη των ε, ε, αρχών αυτών διατησίας. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν ότι υπάρχουν και διαμεθοριακές αρχές διαμεσολάβησης, ότι οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν σε αυτές στην δική τους γλώσσα, στη μητρική τους γλώσσα. Θα πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο, αριθμός τηλεφώνου, email, διαχειδρομική διεύθυνση, οπότε θα γνωρίζει ο καταναλωτές ότι αν υπάρχει κάποια καταγγελία ή κάποια διαφορά, μπορεί, γνωρίζει πού να απευθυνθεί στη χώρα του, στην μητρική του γλώσσα. Και θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα ώστε να γίνεται η διαβίβαση τις υποθέσεις από τη μια χώρα στην άλλη, ας πούμε τη Γερμανία στην Ιταλία και ούτω καθεξής. Διότι θέλουμε να δημιουργηθούν τα πράγματα αυτά και ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι ήδη υπάρχουν πολλές αρχές διαμεσολάβησης στην Ευρώπη που λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο. Γι' αυτό το ερώτημα είναι θα τις χρησιμοποιήσουμε, θα κάνουμε ένα κατάλογο best practices, θα τις αναπτύξουμε ή θα ακολουθήσουμε νέους δρόμους. Το δεύτερο θέμα που θίγει εδώ κατά επανάληψη είναι η ταχύτητα. Δεν έχει νόημα να περιμένει ο καταναλωτη δυο 2-2,5 χρόνια, διότι εκεί δεν αυξάνεται βεβαίω η εμπιστοσύνη. Το τρίτο, χρειαζόμαστε την ανεξαρτησία των ε, αρχών διαιτησία ή των φορέων ε, διαιτησία. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει κάποια εμπιστοσύνη για το που μπορεί να απευθυνθεί να γνωρίζει ότι ο φορέας αυτός θα τον ακούσει και θα τον λάβει σοβαρά υπόψη. Τώρα, αν χρειαζόμαστε υποχρεωτικά την εφαρμογή της εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών, άκουσα ότι στην Ιταλία αυτό συμβαίνει, άκουσα επίσης ότι ο Επίτροπος το σκέφτεται, μπορεί βέβαια, αυτό να είναι αλήθεια. Δεν θα πρέπει επίσης να, η υπόθεση αυτή να συνεπάγεται κόστος σε βάρος του καταναλωτού, διότι εάν γνωρίζει ότι μπορεί πρώτον να χάσει την υπόθεση και δεύτερον να επιβαρυνθεί με το κόστος, ε, δεν θα τολμήσει να προχωρήσει. Ενώ το αντίθετο θέλουμε να του ενθαρρύνουμε. Χρειάζεται και διαμεθοριακός χαρακτήρας, το είπα αυτό ήδη πριν, και κυρίως διαδικασία επιγραμμική. Αυτές είναι κάποιες προτάσεις που ε, προκύπτουν κατά τη γνώμη μου από τη σημερινή συζήτηση όπου κληθήκαμε άλλωστε να υποδείξουμε δρόμους, κατευθύνσεις που μπορούμε να βελτιώσουμε το μηχανισμό αυτό προς το συμφέρον και των παραγωγών. Κυρίω των μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Τα είπε αυτά προηγουμένω και ο Ούγγρο Υπουργό, διότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίε και πέραν τη μεθορίου. Εάν λοιπόν γνωρίζουν τι θα αντιμετωπίσουν εφόσον ας πούμε ε, αποστείλουν ελαττωματικά προϊόντα, Εάν γνωρίζουν λοιπόν τι θα πρέπει να αναμένουν, θα είναι πιο πολύ διατεθειμένες να ε, το πράξουν, να συμμετάσχουν σε τέτοιες, ε, να προσφέρουν δηλαδή τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες, παρά εάν φοβούνται ότι κινδυνεύουν να πέσουν σε περιπέτειες. Άρα θα πρέπει να εξυπηρετούν και οι δύο πλευρές, να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό με όλες τις προτάσεις που σας ενέφερα και πριν διότι μόνο αν υπάρχει υψηλού επίπεδου αποδοχή, μόνο αν ο κόσμος γνωρίζει πού πρέπει να απευθυνθεί, πού μπορεί να απευθυνθεί και ότι θα βρει συνομιλητή ο οποίος θα επιληφθεί τις υποθέσεις τους και θα την προωθήσει, μόνο τότε θα έχουν και τη διάθεση πραγματικά να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καταρχάς ε, συμφωνώ ασφαλώς με τα σχόλια που κάνατε σε ό,τι αφορά τα θέματα εμπιστοσύνης, η διαθεσιμότητα, το αίσθημα ότι οτιδήποτε και να πάει στραβά μπορεί να διορθωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο εκείνο που εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει κάποια διαμεθοριακή συναλλαγή. Όσοι διαβάσατε την πρόσφατη έκδοση του σχετικού scoreboard θα δείτε ότι δεν αναπτύσσεται το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, αναπτύσσεται πάρα πολύ το εσωτερικό, το εγχώριο διαδικτυακό εμπόριο. Το καλό είναι ότι όταν ο κόσμος ε, ξεκινάει και κάνει μια αγορά μέσω του ίντερνετ διαμεθοριακά, αποκτά εμπιστοσύνη σταδιακά και επαναλαμβάνει τις ε, αγορές αυτές. Αλλά είναι σημαντικό το αίσθημα ότι σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά μπορεί να βρει κανείς βοήθεια. Νομίζω ότι αυξάνοντας και τις διαθέσιμα συστήματα ADR, σε τελική ανάλυση δεν σημαίνει ότι θα αποτανθούν πιο πολλά άτομα σε υπηρεσίες ADR απαραίτητα. Θα πρέπει να είναι γρήγορες διαδικασίες και χαμηλού κόστους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας. Άρα η διαθεσιμότητα και η διάθεση ADR θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ε, υπηρεσίες μετά την πώληση και επίσης τελικά αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα αντιλαμβάνονται καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, τα προβλήματα στις υπηρεσίες που παρέχουν και τελικά όλα αυτά θα καταλήξουν στην άλλη άκρη της και πάλι και πιστεύουμε από τις μελέτες μας ότι μέχρι και 4% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ δεν ε, κατανέμονται όπου θα έπρεπε. Και αυτό πλήττει τους καταναλωτές, γιατί τελικά οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν καλές υπηρεσίες δεν απολαμβάνουν τα, ε, τα αναγνωστικά πλεονεκτήματα που θα έπρεπε. Άρα αυτό απασχολεί εξίσου και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Και τώρα να δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, τον Πίτερ Μόρκενς, ο οποίος είναι επικεφαλής και τον είχα προειδοποιήσει ότι δεν θα μπορέσω <laughs> να προφέρω τη λέξη της ε, Ολλανδικής Αρχής ε, που είναι αρμόδια για την ε, ε, διαχείριση του πολύ αποτελεσματικού Ολλανδικού ε, συστήματος διευθέτησης διαφορών. Και νομίζω ότι έχει διαφάνειες. Η κυρία Ρία Όμον Ράιτεν, νομίζω ότι είναι πρόεδρος της ομάδας αυτής, ναι. Σωστά τα λέτε. Καλώ ορίσατε, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μας προφέρετε τη λέξη. Ναι. Τέχεσχύλε κομίσεις. Όπως και το όνομά μου, Ράιτεν, συχνά προφέρεται λάθος. Ε, και αυτή η λέξη είναι δύσκολη. De Geschillen Commissie. Αλλά λειτουργεί άψογα στην Ολλανδία. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω σύντομα την οργάνωσή μας. Αυτό τι σημαίνει. Θα ήθελα να σας ε, πω από τι αποτελείται η Ένωση Οργανώσεών μας. Μετά να σας μιλήσω για το πώς λειτουργούν οι Επιτροπές ε, ε, Διευθέτησης Διαφορών. Θα σας πω ε, την ηλεκτρονική μας διαδικασία, θα σας παρουσιάσω και θα καταλήξω σε συμπεράσματα. Η Ένωση Οργανώσεων μας υπό την Επιτροπή Διευθέτησης Διαφορών υπάρχονται 50 ε, τομεακές οργανώσεις και η οργάνωσή μας ε, βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνες είναι οι οργανώσεις καταναλωτών. Οι οργανώσεις καταναλωτών θέλουν ε, εύκολη και γρήγορη διευθέτηση διαφορών μέσω μια θηρίδα για τον καταναλωτή. Δεύτερος πυλώνας οι επιχειρήσεις που βασικό στόχο έχουν ε, την ε, εξασφάλιση της ποιότητας και τρίτος πυλώνας η κυβέρνηση, η οποία επιθυμεί πέρα από τα δικαστήρια να υπάρχουν και άλλοι πιο εύκολοι και γρήγοροι τρόποι αντιευθέτησης. Ε, βασιζόμαστε σε αυτορύθμιση, δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξης για τους επιχειρήσεις. Όσες θέλουν εθελοντικά εντάσσονται στην Ένωσή μας. Η Επιτροπή διαφορών αναπτύσσεται και μεγαλώνει με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Από το 2005 μέχρι το 2010 έχουν προσταθεί 20 επιτροπές διευθέτησης διαφορών, πάρα πολλέ. Και αυτό καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις ε, αφιερώνουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ποιότητας και θέλουν ασφάλεια για τον καταναλωτή. Στην επόμενη σελίδα βλέπετε τις 50 επιτροπές διευθέτησης διαφορών και στην επόμενη σελίδα σας τα έβαλα με μικρή γραμματοσυρά για να, μην, για να χωρέσουν όλες οι επιτροπές και καλύπτουν σχεδόν όλους τους κλάδους της, ε, των επιχειρήσεων όπου υπάρχουν συναλλαγές. Να σας δώσω κάποιες παραδείγματα. Επικοινωνίας, μάλλον επιτροπές που σχετίζονται με επιχειρήσεις επικοινωνιών και αυτό περιλαμβάνει και τους παρόχους υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Οι επόμενες επιτροπές δραστηριοποιούνται στις οικοδομές, 8-9 περίπου στον αριθμό. Επόμενος κλάδος οι μεταφορές και ιδιαίτερα έχουμε την Επιτροπή για την Αεροπορία η οποία εντάσσεται στις Επιτροπές ε, για τις μεταφορές, η οποία λειτουργεί εδώ και 1,5 έτος και ε, οι επιβάτες, ε, οι καταναλωτέ που έχουν ε, αγοράσει ένα εισιτήριο μπορούν να καταφύγουν, να προσφύγουν στην Επιτροπή αυτή για τυχόν καταγγελίες. Έχουμε και διάφορες επιτροπές που ασχολούνται με θέματα αναψυχής, όπω τα ταξίδια και μία τελευταία που θα ήθελα να σα αναφέρω είναι οι επιτροπέ που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, νοσοκομεία, περίθαλψη κατοίκων. Από τι αποτελείται ε, μια τέτοια επιτροπή. Από τρία ανεξάρτητα μέλη. Η Επιτροπή λοιπόν είναι τελείως ομερόληπτη και ανεξάρτητη. Ακολουθούμε και το σουηδικό μοντέλο. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να κινηθεί εξοδικαστικά ή δικαστικά εάν ε, επιλέξει την Επιτροπή Διαθέτησης Διαφορών υποχρεούνται να την ακολουθήσει και ο επιχειρηματίας. Και επίσης αναγνωρίζονται οι επιτροπές μας αυτές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και πληρούν τους όρους ε, σχετικού κανονισμού σχετικής οδηγίας του 98 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ένα πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο σημαίνει ότι ο Επίτροπος μπορεί να καταγγείλει ψηφιακά και επίσης μπορεί να παρακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια της καταγγελίας σε ποιο στάδιο βρίσκεται η καταγγελία. Μπορεί να ξέρει λοιπόν ανά πάσα στιγμή ο καταναλωτής που βρίσκεται η καταγγελία του. Η ηλεκτρονική είναι η διαχείριση του συστήματος. Υπάρχει ένα μητρό που περιλαμβάνει όλους τους, ε, όλες τις επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική μορφή ε, και όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και βλέπουμε ότι τελικά οι καταγγελίες έχουν αποτέλεσμα έχουν ως ε, αποτέλεσμα την ε, αύξηση της ποιότητας των επιχειρήσεων. Εδώ πέρα βλέπετε στην επόμενη σελίδα κάποια αριθμητικά στοιχεία. Περίπου 10.000 έως 11.000 καταγγελίες επεξεργαζόμαστε κάθε χρόνο. Βλέπετε ότι έχουμε και ένα website, μία ιστοσελίδα. Τέσσερις εβδομάδες κατά μέσο όρο ε, παίρνει η διαδικασία για τον καταναλωτή, για την επιχείρηση και τέσσερις εβδομάδες ε, ακόμα για να εξετάσουμε το σύστημα, το, το, την καταγγελία και τέσσερις εβδομάδες μέχρι να εκδοθεί η απόφαση. Ποιος πληρώνει τώρα το σύστημα αυτό καταρχάς η κυβέρνηση ε, δίνει ένα σταθερό ποσό κάθε χρόνο για τις υποδομές. Οι επιχειρήσεις ε, πληρώνουν το κόστος ε, διαχείρισης όλων των επιχειρήσεων, όλων των υποθέσεων, όλων των καταγγελιών. Όσο πιο λίγες είναι οι καταγγελίες, όσο πιο μικρό είναι το κόστος και ο καταναλωτής καταβάλει 25 έως 125 ευρώ για κάθε καταγγελία και τίποτε παραπάνω, ούτε ευρώ παραπάνω και αν ε, δικαιωθεί ο καταναλωτής του επιστρέφονται και όλα τα χρήματα αυτά. Συμπέρασμα, νομίζω ότι έχουμε ένα πραγματικά μοναδικό σύστημα με, αυτό ε, με την ένωση ε, τέτοιων επιτροπών υψηλής ποιότητας, αξιόπιστο, ενιαίας και εύκολης πρόσβασης, γρήγορο και φθηνό. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια βέλτιστη πρακτική που καταδεικνύει την δέσμευση των κυβερνήσεων, των οργανώσεων καταναλωτών και της, ε, των επιχειρήσεων. Very, Ευχαριστώ πράγματι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να επαναληφθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι ένα παράδειγμα μιας άριστης ε, πρακτικής. Και έτσι τώρα ερχόμαστε τελευταίο ομιλητή, πριν ξεκινήσει η συζήτηση, ο κ. Πιγκάντολης, επικεφαλής της ομάδας καταναλωτών της ΟΚΕ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που είναι ένα άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οθέτησε Επιτροπή του γνωμοδότηση για την ε, ενιαία πράξη σήμερα το πρωί, που και εκεί υπάρχει αναφορά στο ADR, άρα θα μας πει ποια είναι η άποψη της ΟΚΕ για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία μου, τα, τα, πέντε λεπτά ε, δεν με επιτρέπουν να χαιρετήσω όπως αρμόζει αυτή η πρωτοβουλία. Αλλά επειδή είμαι ο τελευταίος του πάνελ, ε, είναι ότι όλα σχεδόν έχουν ε, υποθεί, οπότε θα μπω κατευθείαν επιγραμματικά στο θέμα. Επιτρέψτε μου, κυρία μου, να απαντήσω στον κύριο Malcolm Harbour, που ρώτησε ποια είναι η θέση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δεν επελήφθη στη γνωμοδότησή της ε, των δύο θεμάτων. Άρα η άποψη που εκφράζω τώρα είναι αποκλειστικά προσωπική. Όπως είπατε όμως κυρία μου, χτες μόλις, νομίζω χτες, η ΟΚΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση για την Single Market Act που ουσιαστικά λέμε ότι η προσφυγή δικαιοσύνη είναι ουσιαστικό στοιχείο για να έχει εμπιστοσύνη η αγορά. Ο καταναλωτή, ο συντονισμό, οι, συνομιλίε τώρα όσον αφορά τη συλλογική προσφυγή, τι διάφορα είδη προσφυγή πρέπει να βασίζονται επί νομοθετικών προτάσεων και χαιρόμαστε διότι στο πρόγραμμα εργασιών 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι θα κάνει πρόταση ε, νομοθετική για εξοδικαστική επίλυση των διαφορών και θα κάνει σχετικέ προτάσει. Ε, λοιπόν, ελλείψη χρόνου. Ε, πρέπει να πω ότι πολλές εκφρα... Ε, απόψεις εκφράστηκαν όσον αφορά το θέμα ήδη. Ε, στο... Λοιπόν, Λοιπόν, αναφέρθηκα σε αυτά που θα πω στο τέλος εσαιρετικά τώρα, τέλος πάντων. Έκανα ένα προθύστερο. Λοιπόν, στη συζήτηση πρέπει να δούμε τα δύο, τα δύο θέματα συμπροματικά. Να επιθυμίσουμε όμως σημαντικά έγγραφα Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρχάς, πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απρίλιο 2002. Συστάσεις του, Επιτροπή Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και κάποιε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απόφαση Κλάρο, Λασινή, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Φίλιπς κατά Ελλάδος, που είναι πολύ σημαντικά σημαντικές υποθέσεις. Λοιπόν, ε, όπως είπε και η κυρία Φέντερσπιλ, που ήταν ένας από τους τρεις σωματιφύλακες όπως αποκαλούνται, που ετοίμασε μια γνωμοδότηση της ηγητές για την Single Market Arc. Μια γνωμοδότηση της ηγητές. Αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε με ηρεμία το θέμα. Και δεν θα πρέπει τα ADR να τα συγκρίνουμε με άλλους τρόπους επιλύσεως των διαφορών. Η επίλυση των διαφορών ε, δεν είναι θέμα δικαστικό. Η δικαιοσύνη, απόδοση δικαιοσύνης ανήκει στα δικαστήρια. Μόνο τα δικαστήρια μπορούν να αποδώσουν δικαιοσύνη. Τα ADR είναι ένα έξοχο μέσο επιλύσεως διαφορών. Κυρίως στον τομέα της καταναλώσεως. Αντί να μιλάμε για εναλλακτικά μέσα, θα έπρεπε να λέμε επαρκή μέσα, ενδεδειγμένα μέσα επιλύσεως των διαφορών. Για να κρατήσουμε το A στα αγγλικά το alternative. Λοιπόν, δεν αντικαθίσταται δικαστήρια από αυτά τα μέσα, τα ADR. Είναι συμπλήρωμα χρήσιμο και ίσως αναγκαίο συμπληρώνουν τα δικαστήρια. Λοιπόν, αναφέρθηκαν οι λόγοι χρειάζονται αυτά τα μέσα, είναι, υπάρχει ευελιξία, είναι κοντά στον καταναλωτή, δημιουργεί εμπιστοσύνη, επιλύονται διαφορές γρήγορα, είναι απλή διαδικασία κλπ. Εμπιστευτικός χαρακτήρας, είμαι υπέρ της εμπιστευτικότητας. Για να έχουν πραγματικά εναλλακτικό μέσο επιλύσεως των διαφορών χρειάζεται εμπιστευτικότητα. Υπό προϋποθέσεις, προσχώρηση εθελοντική, ανεξαρτησία Ισοτιμία των μερών. Επαρκής κατάρτιση των διαμεσολαβητών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεσμευτικός χαρακτήρας και εκτελεστικός, εκτελέσιμος χαρακτήρας των αποφάσεων. Αναστολή λοιπόν και του χρόνου παραγραφής. Όσο εξετάζεται το θέμα. Ο Ούγγρος υπουργό είπε και συμφωνώ ότι τα εμπλεκόμενα μέρη των κρατών μελών εν πρώτης πρέπει να αποφασίζουν το σύστημα EDR που είναι το δέον και αναγκαίο. Και το σύστημα είναι bottom-up όπως λέμε. Εκ το κάτω προς τα άνω. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να κάνουμε κάτι σε κοινοτικό επίπεδο. Η απάντησή μου είναι ναι, αλλά. Πρώτα απ' όλα το αλλά. Είπαμε εδώ ήδη κάτι. Η επικουρικότητα, η αναλογικότητα είναι δύο κριτήρια που θα πρέπει να τα αναλύσουμε εις βάθος όταν πρέπει να κάνουμε κάτι στο θέμα σε κοινοτικό επίπεδο. Μετά το ναι. Γιατί? Πρώτα απ' όλα για να εγγυηθούμε μία βάση αξιοπιστίας των ADR σε όλα τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση ότι τα υπάρχοντα ADR σέβονται παραμέτρους προκαθορισμένες και σαφούς. Ποιες παραμέτρους? ανεξαρτησία, αμεροληψία. Κάναμε διάκριση μεταξύ των δύο εδώ. Εγώ δεν μπορώ να διακρίνω τα δύο, τέλος πάντων. Διαφάνεια. Η αρχή της αντιπαράθεσης, αποτελεσματικότητα, ισοτιμία, ισότητα, ελευθερία, εκπροσώπηση, αντιπροσωπευτικότητα, όλες αυτές οι παράμετροι συμπεριλαμβάνονται στις τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98 2001. Αυτά μπορούμε να τα πάρουμε. Τις συστάσεις να τις μεταμορφώσουμε σε οδηγία. Αυτό προτείνω λοιπόν. Οδηγία. Να. Οδηγία. Με τι. Θεμελιώδεις αρχές. Θεμελιώδεις διαδικαστικούς κανόνες. Υποχρέωση ενημέρωση με τη σύναψη των σύμβασης και εντό τη συμβάσεω, μεγάλο περιθώριο πρωτοβουλία των εμπλεκομένων μερών και των κατών μελών, συνεργασία αυξημένη στα πλαίσια του κανονισμού 2006-2004 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει αυτό, κάνει ένα διατύπωση του κειμένου, άρα είναι πολύ καλή ευκαιρία να κάνει κάτι παραπάνω από απλή αναδιατύπωση. Αυτή είναι η άποψη της ΟΚΕ. Το επεξεργαζόμαστε και θα το διατυπώσουμε σε γνωμοδότηση για δημιουργία ενός δικτύου online πάρα πολύ σημαντικό στο διαδίκτυο. Έχω κάποια σχόλια όσον αφορά τις συλλογικέ προσφυγές. Είχα να πω κάτι την ιδιαιτερότητα αυτή, δεν θα το πω, δεν έχω χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ιδού τα όρια που έχουμε δεν ξέρω αν έχουμε μείνει πολύ πίσω στην προσπάθειά μας ή αν μπορούμε να κάνουμε κάτι έγκαιρα και να πετύχουμε τα, τα αποτελέσματα. Εντάξει. Καλό τέλος στην παρέμβασή σας. Όλοι έχετε δυνατότητα να πάρετε το λόγο. Σκοπός της συζητήσεως τώρα είναι να κοιτάμε προς το μέλλον. Όχι να δούμε τι ήδη υπάρχει, και να κάνουμε τέτοια απογραφή. Όσοι έχετε ιδέες για το μελλοντική, τη μελλοντική μορφή νομοθετικής προτάσεως, ας μας μιλήσετε. Πείτε το μας. Πολλοί έχουν ιδέες. Μάλκομ, Καρλάιλ, η κυρία εκεί κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ σήμερα. Θα ήθελα καταρχάς να επενέσω την πρωτοβουλία του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νομίζω ότι κάποια από τα βασικά ζητήματα είναι κοινά. Όλοι συμφωνούμε για την πληροφόρηση. Νομίζω ότι τρεις φορείς εμπλέκονται οι κυβερνήσεις που θα πρέπει να τηρούν ένα μητρό των ε, συστημάτων που υφίστανται στην επικράτειά τους. Οι επιχειρήσεις επίσης θα πρέπει σαφώς να ενθαρρύνονται για να συστήσουν τέτοια συστήματα και να ενημερώνουν το κοινό. Και νομίζω ότι καλή ιδέα θα ήταν να υπάρχει και ένας αυστηρός κανόνας για τον οποίο, ο οποίος θα προβλέπει ότι οι δικηγόροι θα πρέπει να συστήνουν στους πελάτες τους αυστηρός να καταφεύγουν σε μεθόδους ε, διαμεσολάβησης πρωτού καταφύγουν στο δικαστήριο, γιατί το δικαστήριο είναι και πολύ ακριβό. <coughs> Δεύτερο σημείο που ήθελα να θέσω περί αξιοπιστίας. Προκειμένου να υπάρχει αξιοπιστία στα συστήματα αυτά, είναι πολύ επιθυμητό να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και να είναι πιστοποιημένα τα συστήματα με βάση τα κριτήρια αυτή. Ακούσαμε και στην Ολλανδία τι γίνεται, υπάρχουν σχετικά τέτοια συστήματα στον Εμένο Βασίλειο και παντού και σε πολλές άλλες χώρες. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, αυτό θα βελτιώσει την αξιοπιστία. Τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η εθελοντική, ο εθελοντικό χαρακτήρα ε, των συστημάτων διευθέτηση διαφορών. Δεν μπορούμε να το υπαγορεύσουμε αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά βασικό. Γιατί αν κινηθούμε προς υποχρεωτικό ADR, νομίζω ότι θα καταστρέψουμε τον ίδιο το σκοπό του συστήματος. Τελευταίο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να θεωρεί τα δικαστηρία όχι μόνο ως ε, ένα σύστημα για την εκδίκαση υποθέσεων, αλλά και ως ένα σύστημα για την υποστήριξη του ADR. Νομίζω και σκέφτομαι το Ολλανδικό παράδειγμα όπου το δικαστήριο ουσιαστικά επιβλέπει τις διαδικασίες διαμεσολάβησης για να διασφαλίσει τους δίκαιους όρους και να διασφαλίσει ότι αν τα μέρη το επιθυμούν το δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφαση διαμεσολαβητή και την καθαριστά νομικά δεσμευτική και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο θέμα της δικαστικής επικύρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όπως μου υπενθύμησε ο Μάλκομ και έπρεπε να το είχα πει στην αρχή, θα σας παρακαλούσα να είσαστε σύντομοι και λακωνικοί στις εισηγήσεις σας. Δύο λεπτά. Θα ζητήσω από τους επόμενους ομιλητές να είναι το συντομότερο το πιο σύντομοι πιο Και επίση παρακαλώ να, συστη... μας πείτε ποιο είστε, ποια είστε. Από τη Σλοβενία είμαι και είμαι δικηγόρος και είμαι επίση διαμεσολαβητή στο Περιφερειακό Δικαστήριο στην Λουμπλιάνα, αλλά συμμετέχω εδώ ως ε, δικηγόρο σε θέματα καταναλωτή και θα ήθελα να συνεχίσω στα Σλοβενικά, αν γίνεται. Ε, το συστήματα ADR σημειώθηκε ότι θα πρέπει να είναι δίκαια προς τους καταναλωτές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Και επίσης αυτό σημαίνει ότι οι ενώσεις καταναλωτών θα μπορούν να αγγιηθούν για τα συστήματα αυτά και το ίδιο ισχύει και για τους δικηγόρους προκειμένου τα συστήματα ADR να είναι αξιόπιστα θα πρέπει να είναι σωστές, δίκαιες και αμερόληπτες ε, οι αποφάσεις που λαμβάνουν και ως εκ τούτου ο κάθε διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι να, γνωρίζει τις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε υπόθεσης. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο η διαμεσολάβηση. Το θέμα είναι ότι η λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τις ε, διαφορές καταναλωτών καταναλωτικής φύσης είναι διαφορετική φύσης. Είναι διαφορετική φύση από όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ δύο επιχειρήσεων. Είναι συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά των ε, διαφορών που εμπλέκουν και καταναλωτές. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη κατά την κατάρτιση των κοινών ε, αρχών για τη διαμόρφωση των συστημάτων ADR. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα και του απορρίτου της εμπιστευτικότητας, που αποτελεί και τη βάση των διαδικασιών ε, διευθέτησης διαφορών. Αυτό δεν είναι πάντα θετικό για του καταναλωτέ και εδώ πέρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί οι ε, διαφορές ε, που εμπλέκουν καταναλωτέ εμπλέκουν πολλά μέρη σε πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο θέμα καταναλωτή και επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις τα θυγόμενα μέρη είναι πιο πολλά στον αριθμό. Και αυτό θα πρέπει να το συνδέουμε και με τις αιτήσει εκθέσεις ε, για τα χαρακτηριστικά των ε, διαφορών που διευθετούνται σε, ένα, σε μια οργάνωση ADR προκειμένου αυτό να ωφελήσει και άλλους καταναλωτές, προκειμένου να αποφύγουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές και προκειμένου να λάβουν τέρμα κακές πρακτικές από πλευρά των επιχειρήσεων. Και έτσι μπορούμε να ενθαρρύνουμε και τον δικαιό ανταγωνισμό στην αγορά, γιατί πάντα λαμβάνουμε αποφάσεις σε ό,τι αφορά παραβιάσεις. Οι επιχειρήσεις... Κάποιες επιχειρήσεις όμως ποτέ δεν είναι αντίθετες, μάλιστα λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος στο έδραν 79. Γεια σας, καλησπέρα. Βίντσαντ Νίλμεντ από, την... από τα εμπορικά επιμελητήρια, από Ένωση Εμπορικών Επιμελητηρίων. Να απαντήσω σε κάτι που έχει θυχτεί επαναλημμένα. Νομίζω ότι είναι αρκετά απλοϊκό να πιστεύουμε ότι το ADR είναι φθηνό. Ποτέ δεν είναι φθηνό, καταρχάς. Και να σας πω ότι πριν από κάποια χρόνια ιδρύσαμε ένα επιγραμμικό τέτοιο σύστημα καταγγελίων και αν θέλουμε να είναι ποιοτικό το σύστημα αυτό χρειάζονται εμπειρογνώμονες, ε, χρειαζόμαστε γραμματεία, χρειαζόμαστε κάποια συστήματα διαχείρισης ποιότητας και όλα αυτά σημαίνουν κόστος. Και αυτό το κόστος συχνά δεν ανακτάται από τα μέρη όταν είναι πιο υψηλό το κόστος της ε, διένεξης, της διαφοράς. Ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται και διαμαθεωριακό χαρακτήρας. Θα με ενδιαφέρει η περαιτέρω αξιολόγηση του σύνδεσης μεταξύ της ποιότητα και του κόστους ενός τέτοιου συστήματο διευθέτησης διαφορών. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ω τώρα. Και πώς μπορούμε να βρούμε ένα σύστημα χρηματοδότησης για κάποιες διαφορές χαμηλού χαμηλής αξίας και κάποια συστήματα από ό,τι κατάλαβα είναι χρηματοδοτούμενα από δημόσιες δαπάνες. Υπάρχουν άρα για να ρωτιέμαι ιδιωτικά τέτοια ιδιωτική χρηματοδότηση στον τομέα αυτό και μήπως υπάρχουν και κάποιες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μάλιστα. Και τώρα λέει η πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ από το Πανεπιστήμιο του Oxford, της Εξφόρδης. Κάνουμε έρευνα και θέλω να αναφερθώ στο θέμα της τεχνικής. Οι δομές και αρχιτεκτονική κάποιων φορέων ADR ποικίλουν πάρα πολύ μεταξύ χωρών. Οι τεχνικές όμω που χρησιμοποιούν είναι πολύ παρόμοιε όσον αφορά τη μεσολάβηση. Όταν είδαμε τα καλύτερα παραδείγματα, τι βλέπουμε. Κάποια αλληλουχία τεχνικών, δηλαδή διαπραγματεύσει μεταξύ μερών, συνδιαλλαγή, διαμεσολάβηση μετά ακολουθεί από κάποιο εμπειρογνώμονο, Μετά δεσμευτική διαιτησία που απαιτεί μεγαλύτερη εξαρτησία ή το δικαστήριο και πολύ συχνά το δικαστήριο είναι τελευταίο και είναι η απειλή του δικαστηρίου που βοηθά να λειτουργήσει το ADR. Τα επόμενα δύο σημεία που έχω να αναφέρω σχετίζονται με το πρόβλημα της έλλειψης ορατότητας, έλλειψης χρήσεως, έλλειψης υποστήριξης ε, υπογραφή συμμετοχής και καλύψεως τομέων. Δύο πράγματα, δύο στοιχεία μπορούν να μεταμορφώσουν την ολικόνα εικόνα. Πρώτον, ενιαία αγίδα, ενιαίο πλαίσιο, αυτό που έκανε η Ολλανδία. Και κάποιες σκανδιναβικές χώρες βρήκαν παρόμοια λύση. Την απάντηση την έχουν η Ολλανδία. Να ξέρουν και επιχειρήσεις και οι καταναλωτές ότι υπάρχει Συμβούλιο Φορέας για την Διαφορών και αυτό επιλύει τη διαφορά που έχουν διάφορε χώρε, διαφορετική διαμοσολαβητή, διαφορετικά σχήματα, διαφορετικοί μηχανισμοί, διαφορετική δια... Αν ξέρετε ότι κάτι υπάρχει, αν ξέρετε πώ αποκαλείται, τότε λειτουργεί το σύστημα. Και ο κόσμο ενδιαφέρεται περισσότερο να δημιουργεί κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει ένα ενίο συγκεκριμένο ποιοτικό πλαίσιο. Τρίτον, συχνά το ADR το θεωρούμε σε συνάρτηση με τα δικαστήρια. Εάν βάλουμε και ρυθμίσεις και νομοθεσία, τώρα τι έχουμε ένα εντελώς ποιοτικό σύστημα ανάδρασης που θέλουν επιχειρήσεις. Δεν επιλύεται μόνο η διαφορά, συλλέγονται πληροφορίες με το σύστημα υποβολής διαμαρτυριών και καταγγελιών και τα αποτελέσματα των, της επιδιατησίας και των δικαστηρίων και τροφοδοτείται από τους φορείς ρύθμισης αυτορύθμισης και βελτιώνεται η ποιότητα μέσω της ανάδρασης και προωθεί τη χρήση του ADR και ταυτόχρονα και την ποιότητα της αγοράς εργασίας. Και αν το κάνετε αυτό, η Ρίστο εν παρόδο ε, έχετε ε, κάνει πολλά πράγματα για να βελτιώσετε την επίλυση διαφορών μέσω συλλογικής ε, προσφυγής. Η κυρία έχει το λόγο. Thank you very much. My name is Antje Federke and I'm Secretary General of the International Association of Legal Expenses Insurance. Um, I first... Είμαι γενική γραμματεύσει. Κοιτάξτε, αυτή η διαβούλευση είναι πάρα πολύ ευρεία. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικά συστήματα, μεθόδους, μηχανισμούς. Οι μέθοδοι ίσως ε, είναι παρόμοιες εντός διαφορετικών ADR. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επενθυμίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να έχει σαφείς ορισμούς, να υπάρχει βεβαιότης του τι συζητείτε. Και έρχομαι σε κάτι άλλο τώρα. Προαπαιτούμενα ίσως να ποικίλουν για τα διάφορα συστήματα. Μιλούσαμε το χάρη για εμπιστευτικότητα, μιλούσαμε για δημοσίευση των αποφάσεων για τη διαμεσολάβηση παραδείγματι είναι πολύ σημαντικό να επικρατεί και να γίνεται σεβαστή η εμπιστευτικό Αλλιώς δεν θα επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα από τη διαμεσολάβηση. Εφόσον μιλάμε για το μέλλον, θα ήθελα να φέρω στην εικόνα και την ασφάλιση νομικής προστασίας. Την ασφάλιση νομικής προστασίας σε πολλές χώρες οι ασφαλιστές κοιτάνε τι δυνατότητες υπάρχουν στα πλαίσια της διαμεσολάβησης. Είμαστε στην αρχή της Τρία στοιχεία μπορεί να, να βοηθηθούν από την ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα ευαισθητοποίηση. Αν είναι κατάλληλη υπόθεση, οι ασφαλιστές εξασφαλίζουν ότι οι ασφαλισμένοι θα γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα σύστημα IDR τα κενά μετά που υπάρχουν. Θα εκαλύπτονται όλες οι διαφορές ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσεως. Τέλος, εξίσου σημαντικό, κόστος. Τα ασφάλιστρα των ασφαλισμένων θα εκάλυπταν και το κόστος της ε, διαμεσολαβήσεως. Άρα υπάρχει κάποιο περιθώριο ε, για μας, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιζομένους ε, για να καλύπτεται αυτή η διαμεσολάβηση. Δύο τελευταίες παρεμβάσεις για να δώσω χρόνο στους ομιλητές να απαντήσουν. Πολλοί ζητάνε το λόγο, πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο. Ζητούν πολύ το λόγο. Ένας εδώ, ένας εκεί, εκεί, εκεί. Λοιπόν, τέσσερις. Παρακαλώ να είσαστε πάρα πολύ σύντομοι. Ένα λεπτό ο καθένας. Γκρέαμ. Ε, Τρία σύντομα σχόλια πρακτικού χαρακτήρα για τα διαμεθοριακά. Συμφωνώ με τον Chris Hodges ότι ο μηχανισμός εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ε, αγωγών αποζημιώσεων. Δεύτερο, για διαμεθοριακές υποθέσεις, όντως οι καταναλωτέ πρέπει να γνωρίζουν σε ποιον θα απευθυνθούν. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας σε κάθε χώρα μέλος και μπορεί <clears throat> να υπάρχει και, μια διαδικασία διαβίβαση των υποθέσεων από ένα σημείο επαφή σε άλλο. Τρίτο, εμπιστοσύνη στα συστήματα ADR που πρέπει να παρακολουθούνται για την συμμόρφωσή τους με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και βεβαίω να υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση. Και το ADR να ξεκινά στην χώρα του καταναλωτού και σύμφωνα με τους κανόνες της. Τέλος, οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε ένα νομικό πλαίσιο και να λαμβάνουν υπόψη τα ε, θέμητα ε, των καταναλωτών. Μάλιστα, να περιστείτε σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Γιολάντα Κέσα διευθύντρια του ECC Σουηδίας. Πάλι για το αμοιβαίως επωφελέ. Το σύστημά μα λειτουργεί στην Σουηδία καλά. Και πολλέ πολλές επιχειρήσεις πώληση για παράδειγμα αυτοκινήτων συμμετέχουν στο ADR και το προσφέρουν και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο γιατί είναι και ένα μέτρο αποκατάσταση εμπιστοσύνης από πλευράς καταναλωτών και ιδίως εφόσον γίνεται και διαμεθοριακά εν, εντείνεται ο χαρακτήρας αυτός του αμοιβαία υποφελούς. Σας ευχαριστώ. Εσείς κύριε. Το τέστα ΣΑ, Κόνιγκ. Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών, κάποιες σκέψεις να εκφράσω. Πρώτα, οι δύο συστάσεις. Υπάρχουν ασυνέπειες που ήδη τονίστηκαν. Διαφάνεια σημαντικότατη για τον καταναλωτή. Εμπιστευτικότητα όμω. Αντίφαση μεταξύ νομιμότητα και ισότιμη προσέγγισης. Άρα θα πρέπει οι ασυνέπειες να αφαιρεθούν. Να υπάρχει ένα κείμενο, μια οδηγία που καλύπτει τις δύο συστάσεις. Δεύτερο σχόλιο σχετικά με την ε, χρησιμότητα ευρωπαϊκού κανονισμού για ε, τα μικρά προβλήματα, εκεί ίσως μπορούμε να βρούμε στοιχεία που μπορούν να σωματωθούν σε ένα EDR. Το πρόβλημα της μετάφρασης. Υπάρχουν τυπικά έντυπα που μπορούν να μεταφραστούν ως έχουν, μετά ότι δεν υπάρχουν σημικές υποθέσεις, δεν υπάρχουν, ε, δικα, δεν ε, δικηγόροι, ε, δεν, οι δικαστές ας πούμε επιχειρηματολογούν. Συμφωνώ με αυτό που είπε η Μόνικα Κρόιζα. Πρέπει να έχουμε ένα template, μια βάση, μια μορφή ε, τυπικού τύπου για την ε, μορφή του συστήματος για τη μεσολάβηση ε, και η διαφάνεια μετά σημαντική, όχι μόνο όσον αφορά την ύπαρξη του συστήματος αλλά και τα αποτελέσματα. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να έχει μια βάση δεδομένων που του δίνει όλα τα αποτελέσματα ενός συστήματος διατησίας Άρα θα έπρεπε επίσης ο καταναλωτής να έχει πληροφορίες ε, για όλες τις δυνατότητε προσφυγή που υπάρχουν. Χρειάζεται ένα πλήρε σύστημα που θα έχει διασύνδεση link με άλλες τις μόνε υποθέσεις για να ενημερώνει το καταναλωτή. Άλλο σχόλιο που αφορά τη διαφάνεια. Νομίζω ότι ε, συστήματα που προβλέπουν μέτρα προληπτικά είναι εξίσου σημαντικά. Πιστεύω ότι η διαφορά μπορεί να αποφευθεί μέσω τυπικών μοντέλων ε, ε, συμβάσεων με ελάχιστε ρήτε, Το Ολλανδικό σύστημα και το Βελγικό σύστημα είναι καλά παραδείγματα. Υπάρχουν τυπικά μορφέ, τυπικέ ε, πρότυπε συμβάσεων που εμπεριέχουν στοιχεία που αφορούν την ενημέρωση και την πρόληψη που είναι πολύ καλό γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ένας τελευταίος ο κύριος εκεί και ζητώ συγγνώμη από όσους τυχόν απογοητεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φερνάντε Ντελαρόσα, Πανεπιστήμιο τη Γρανάδα, καθηγητή διεθνού δικαίου. Με προσεκάλεσαν εδώ ε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της Ισπανίας και θα το γυρίσω τώρα στα Ισπανικά. Λοιπόν, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα όλη η συζήτηση απογευματινή και Πολύ τόσο υπόθηκαν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν νομίζω ότι τονίστηκε αρκετά η σημασία και η αξία των ADR για τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές, στο διασυνοριακό εμπόριο. Αυτό που θέλω εγώ να θίξω είναι το εξής. Συζητάμε την ανάγκη δημιουργίας του καταλήλου πλαισίου που θα επιτρέπει τις δέουσες εξελίξεις. Αλλά αυτό που δεν θα πρέπει να λησμονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα τμήμα του ρόλου που πρέπει να παίξει όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα είναι η προστασία των καταναλωτών. Πολλοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη που υπάρχει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία οδηγία θα τονίζει την προστασία των καταναλωτών μέσω των διαφόρων εικονικών πλατφορμών βάσεων που μας δημιουργεί και επίσης και η οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα πρέπει να, δίνει, να δημιουργεί ένα δίκτυο ασφαλείας νομικό η Ευρώπη. Πώς θα πρέπει να καθορίζει σαφή κριτήρια ώστε οι εταιρείε που παρέχουν υπηρεσίες ε, να έχουν ένα είδος πιστοποίησεως. Αυτό θα έχει πολλές συνέπειες, πρώτα απ' όλα. Θα μπορεί να εμπιστεύεται το σύστημα καταναλωτής. Θα έχει ένα σήμα, ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης αυτό το δίκτυο. Ε, επίσης θα υπάρχουν σχέσεις με τους ομολόγους φορείς των κρατών μελών. θα μπορεί να γίνει διαμεσολάβηση ή επιδιατησία online. Τέτοιο μηχανισμό θα ήθελα να δω να αναπτυχθεί περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο χρόνος προχωρεί. Θα στραφώ τώρα στους αγορητές μας. Αυτό είναι μια πρόσκληση αν θέλετε, αλλά βεβαίως δεν είναι υποχρέωσή σα, αν θέλετε να απαντήσετε. Ας αρχίσουμε τον τελευταίο, τον κύριο Πεγάδο Λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου πολύ σύντομα. Η Κομισιόν βρίσκεται ενώπιν ορισμένων θεμελιωδών επιλογών. Πρώτον, εθελοντικό το σύστημα ή εξαναγκαστό. Την προηγούμενη εβδομάδα στην χώρα μου απεφάσισε η κυβέρνηση να προχωρήσει στην απαραίτητη διαιτησία μονάχα για θέματα θεμελιωδών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό θα ήταν μια λύση αν ήταν βέβαια γενική για όλους. Μια πρώτη επιλογή λοιπόν που θα πρέπει να γίνει. Το άλλο είναι εμπιστευτικό, εμπιστευτικός ή μη χαρακτήρας. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ είμαι υπέρ του εμπιστευτικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε πραγματικούς μηχανισμούς εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών. Και το τρίτο που πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η χρηματοδότηση του κόστους. Ένας από τους παρεμβαίνοντες είπε ότι δεν είναι διόλου δωρεάν το σύστημα. Έχει κόστος. Έχει κόστος λειτουργίας, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο. Πρέπει να δούμε. Είναι ωραία τα συστήματα αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούν να λειτουργούν ορθά, με επάρκεια. Συμφωνώ με έναν από τους προηγούμενους ομιλητές ότι η ποιότητα ασφαλώς είναι πάγεται και κόστος και φαντάζομαι ότι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο έχουμε για παράδειγμα εμείς είναι μεγάλη επένδυση και η κυβέρνηση χρηματοδότησε κατά το ίμιση και οι επιχειρήσεις επίσης αλλά για τον καταναλωτή είναι φτηνό το σύστημα, 25 με 125 ευρώ. Και για, τον, ε, για την κυβέρνηση είναι φτηνό το σύστημα, γιατί αν ο καταναλωτής, κάθε καταναλωτή πήγαινε στο δικαστήριο, το κόστος ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και για τι επιχειρήσει όμω ε, είναι πιο φτηνό το σύστημα, γιατί όσο πιο λίγε είναι οι καταγγελίε, τόσο πιο μικρό είναι το κόστο. και θα πρέπει να το δούμε και στο όλο πλαίσιο τη διαδικασία ε, marketing. Και μια τελευταία παρατήρηση. Τρεις ώρες, ε, ε, μάλλον τρεις ώρες αμοιβή του δικηγόρου είναι το έξοδο που δίνει ο για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το ADR είναι η τελευταία δυνατότητα για γρήγορη και φτηνή επίλυση ε, διαφορών. Δεν είναι φτηνή λύση, αλλά είναι πιο φτηνή από άλλες πιο φθηνή από άλλες διαδικασίες οργανώσεις ε, ε, διατησίας που είναι αξιοσέβεστες αλλά δεν είναι κατάλληλες για την επίλυση τέτοιων διαφορών. Για την Γαλλία, για τη Μέντεφ, θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να πληρώσουν το κόστος της διαμεσολάβησης. Δεν ζητούμε από κανέναν άλλον να μας πληρώσει τα έξοδα. Ο ρόλος μιας ένωσης επιχειρήσεων είναι να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις δεσμεύονται για την ποιότητα του ADR, να δίνουν στον καταναλωτή την εγγύηση της αιμεροληψίας και να διευρύνουν επίσης τον, την τομεακή κάλυψη και γραφική κάλυψη της διαμεσολάβησης. I Πληρώσουμε uh, τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είμαι τελευταίος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής που μιλώ. Ευχαριστώ πλουσιότατη, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον πρόσωπο της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών για τη λήξη των εργασιών. Ευχαριστώ Τζάκη ε, που δίθυνε σε αυτό το τμήμα της συζήτησης. Λοιπόν, εγώ είχα πολύ λιγότερη δουλειά από ό,τι συνήθω. Ε, το απόλαυσα, κράτησα πολλές σημειώσει. έμαθα πολλά πράγματα, συνέλεξα πολλές ιδέες και γι' αυτό χρησιμεύει με τέτοια ακρόαση. Λοιπόν, να πω κάνα δύο σχόλια στο τέλος. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρότεινε αυτή την κοινά οργανωμένη εκδήλωση. Είναι άριστο παράδειγμα συνεργασίας και είναι κάτι που σίγουρα θεωρώ ότι θα θελήσουμε να προωθήσουμε όσο προχωρά αυτή η προσπάθεια. νομίζω ότι η άλλη σκέψη που έχω και θέλω να εκφράσω είναι η εξή. Υπάρχουν πάρα πολλέ γνώσει στον τομέα και θα πρέπει να αντλήσουμε την πηγή τη γνώση και πολλοί από εσά θα ήδη έχετε δώσει τι ιδέε αυτέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπω τόνισε ο Επίτροπο και όπω είπε ο κ. Σέχοβε, για να εκφράσει τα κράτη-μέλη, και οι δύο είπαν λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία προσθέσει αξία σε αυτά που ήδη γίνονται, αλλά θα πρέπει όμως να τλήσουμε από την εμπειρία και να βρούμε όμως με ποιους τρόπους μπορούμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες και ίσως να έχουμε κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι θα αυξήσουν την ποιότητα, θα αναπτύξουμε καλές πρακτικές, δεντολογικούς κώδικες, αλλά σαν Επιτροπή Στασίας του Καταναλωτού στο Κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε, να ασχοληθούμε θέματα διασυνοριακά και να τα βελτιώσουμε. Άρα πρέπει να αυξήσουμε τη συνεργασία των ε, καταναλωτών. Υπάρχουν υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη-μέλη ε, και πολύ συχνά η ομάδα της Τζάκης συνεργάζεται με τους ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα αυτό και σε πολλές περιπτώσεις ε, θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για μας γιατί συνεπάγεται περισσότερους πόρους που θα πρέπει να έρθουν από τα κράτη-μέλη και αυτό είναι ένα συνεχές θέμα που αντιμετωπίζουμε μπροστά μας σε πολλές εργασίες μας όπως υποπτή της αγοράς και άλλους τομείς επίσης όπου θεωρούμε ότι α, θα πρέπει να γίνουν πράγματα άρα πρέπει να το προσέξουμε. Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι και πρέπει να προσέξουμε το θέμα. Τεχνολογία επίσης ε, είναι ο μεγάλος μας φίλος ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε, παραδείγματα κυρίως από τους Ολλανδούς σχετικά με πώς η πληροφορική και τα εργαλεία της χρησιμοποιούνται και περιμένει φράση τα σημεία, η ενιαία θηρίδα, τα ενιαία σημεία, μοναδικά σημεία επαφής, ενιαία σημεία επαφής. Αυτοί που επεξεργάστηκαν την οδηγία υπηρεσιών θα γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζει ένα πρόγραμμα για αυτές τις ενιαίες θηρίδες και επένδυσαν πολύ τα κράτη-μέλη σε online εργαλεία και είναι εργαλεία που προσπαθούν να πλαισιώσουν, να συλλέξουν πληροφορίες και να επιτρέπουν στους συνομιλητές όταν μπαίνουν στο σύστημα να προχωράνε σταδιακά μέσω επιλογών. Άρα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα και αυτά τα εργαλεία υπάρχουν τώρα διαθέσιμα και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που το είπαν αυτό, δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα που θα έχουν οι καταναλωτέ να αντλήσουν από πόρου, να ενημερωθούν και να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουν. Και κάπου ίσω να να υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Να διαλέξουν δηλαδή ένα σύστημα διαμεσολάβησης. Ετέθησαν διάφορα ενδιαφέροντα θέματα για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων. Και οι καλές επιχειρήσεις θέλουν να συμπεριληφθούν σε τέτοιο σύστημα ή τους κάνει καλό στις δουλειές τους. Είναι κάτι καλό και για τους καταναλωτές να μπουν στο σύστημα και πολλές επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση, η αντιμετώπιση προβλήματος του καταναλωτή πολύ συχνά σημαίνει ότι ο καταναλωτή αυτό θα μείνει μαζί σου διαβίου, διότι συμπεριφέρθηκε τόσο καλά και εμείς ήμασταν σε επιχειρήσει. Ε, σε επιχειρήσει ξέρουμε ότι είναι αληθές αυτό το πράγμα. Ένα φίλο μου δούλεψε στον τομέα και μου υπενθύμησε ένας, κάτι, ένα Ιαπωνέζικο ρητό, ελπίζω να τα πάνε καλά τώρα οι Ιαπωνέζοι, και είπε ένα πρόβλημα είναι ένα βουνό με θησαυρού και αν αντιμετωπίσει επιτυχώ με ένα, ένα, ένα πρόβλημα μαθαίνει πολλά. Το θέμα τώρα, εμπιστευτικότητα, διαφάνεια, πώς εξισορροπούνται, όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι σωστό να υπάρχει εμπιστευτικότητα στην επαφή που έχει κατανοτήσει με το σύστημα. Και είναι σημαντικό και το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται και να χρησιμοποιείται με διαφάνεια, διότι ουσιαστικά δημιουργείται νομολογία. Και οι κατανοτές μπορούν να ανακαλύψουν πολλά για την υπόθεσή τους βλέποντας τι έγινε σε παλιές υποθέσεις. Και όσο ε, συσσωρεύονται οι πληροφορίες, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να φτάσει εσύ σε ένα συμπέρασμα, διότι ξέρεις ότι κάποιος είχε αντίστοιχο πρόβλημα με το δικό σου και μπορεί να επιληθεί αρκετά γρήγορα. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες προκλήσεις έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά το έργο τη Επιτροπή, συνεργαζόμαστε στενά με του συναδέλφου τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και μετά χαρά είδε ότι ο κ. ήταν εδώ και Βαντεζάρη, ε, και ο κύριος Λένερ και εγώ ε, συνεργαζόμαστε με την νομική επιτροπή λοιπόν και είναι ένα θέμα για την πολιτική, για τα ADR, ε, νομική πολιτική, τι κάνουμε τους καταναλωτές. Μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλες επιτροπές, το είδαμε, όπως και για την πράξη την ενιαία αγορά θα είστε στην πρωινή μα συνεδρίαση πολλοί από εσά. Θέλουμε να πετύχουμε το ίδιο επίπεδο συνεργασία για θέματα όσον αφορά την εναλλακτική επίλυση διαφορών, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στι ιδέε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είμαι σίγουρο ότι αυτό δεν θα αποτελεί την πρώτη μα ακρόαση, διότι θα θέλουμε να καλέσουμε πολλού από εσά να επανακάμψετε και να έρθετε εδώ και να μα μιλήσετε ξανά για μελλοντικέ προτάσει. Έτσι, αυτά είναι τα τελικά μου σχόλια. Ήταν πολύ πλούσια η όλη εμπειρία. Θα ήθελα, όπω ξέρουν τα μέλη τη Επιτροπής μας, θα το ξαναείδατε, το κάνω αυτό. Σε επενδυμίσω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής αγορά έχει μια, ετοιμάζει μια πολύ έτσι εφημερίδα, έτσι ένα έντυπο, newsletter. Ε, δεν, δεν γράφω εγώ αυτό, το συντάσω εγώ το έγγραφο, έχω μια πολύ καλή ομάδα. Υπάρχει αντίγραφο εκεί, άμα θέλετε πάρτε το. Αλλά θα θέλαμε να παραμείνετε σε επαφή μαζί σα. Και πίσω στη σελίδα βλέπετε, μπορείτε να μπείτε στους, ε, στο δίκτυο των φίλων τη ΣΥΜΚΟ και θα σας έρχεται αυτομάτως ε, ηλεκτρονικά αυτό το έγγραφο. Θέλουμε να φτάσουμε στους, στα 1500 μέλη. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο γι' αυτό και εδώ θα σταματήσω, διότι είναι μια ανακοίνωση αποκλειστική αυτή που κάνω. Δηλαδή, αυτό, αυτός που θα είναι ο χιλιοστός καλείται να γευματίσει μαζί μου στο εστιατόριο των μελών.